Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Καλωσορίσατε για τη διακυβερνοβουλευτική μας ε, συνάντηση της Επιτροπής που εγγράφεται στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας βάσει του άρθρου 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου. ή ε, μάλλον του συμβών για την σταθερότητα, τη σύγκληση και τη διακυβέρνηση, για να είμαστε ακριβέστεροι, και στα πλαίσια της προετοιμασίας της Αρινής ε, Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διπλή λοιπόν η άσκηση αυτή και μας έχει συγκεντρώσει εδώ ε, ως αρμοδίους για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, είτε πρόκειται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Επιτροπή του Κοινοβουλίου ή για την εκάστοτε Επιτροπή της Εθνικής Βουλής. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο αυτή η διάσταση είναι για μας σημαντική στα πλαίσια και στην καρδιά αυτής της διαδικασίας. Και ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι κατά κύριο λόγο αυτό είναι αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών, τα οποία όμως αποφασίζουν για ζητήματα που έχουν πολύ άμεσες επιπτώσεις παντού, σε όλους τους προσανατολισμούς που αποφασίζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε αυτά τα θέματα σε συνεργασία. Για το λόγο αυτό επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλο αυτό το εγχείρημα και η άσκηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κατά κύριο λόγο ε, βλέπει να συνεργάζονται η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, αλλά και η Επιτροπή Προϋπολογισμού, διότι θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να εγγράφονται και αυτά στους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που εκάστοτε χαράσουμε. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ε, θερμότατα τα Εθνικά Κοινοβούλια για τις πάρα πολύ σημαντικές τους συνεισφορές, 12 τον αριθμό, ε, που ε, στάλησαν ως απάντηση στο ερωτηματολόγιο που είχε αποσταλεί και έρχονται αυτές οι απαντήσεις να διαφωτίσουν τις εργασίες μας. Όλα αυτά τα έγγραφα ε, θα είναι στη διάθεσή σας στο διαδίκτυο. Σήμερα ε, διανέμονται σε έντυπη μορφή, θα τα βρείτε στο ίντερνετ ε, ως στοιχεία αναφοράς για να μπορείτε να ανατρέχετε για να διαπιστώνετε τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες. Θα ήθελα να κηρύσω την έναρξη του πρώτου τμήματος των εργασιών μας. Σήμερα το πρωί επιλέξαμε να χωρίσουμε τη συνεδρίαση σε δύο τμήματα. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα αφορά ιδιαίτερα την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, της ΟΝΕ, που μας απασχολεί σφόδρα. Και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω σήμερα στο πάνελ πρώτα ε, σας κύριε Υπουργέ ε, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας της Προεδρεύουσας χώρας ε, της Ελλάδας. Καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Καλημέρα σας. Τώρα πλέον έχουμε γίνει φίλοι σχεδόν. Έχουμε άλλη μια φορά να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και χαίρο γι' αυτό. Επίσης καλωσορίζω θερμότατα τον κύριο Δημήτρη Κρεμαστινό, πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Βουλής των Ελλήνων ε, που επίσης θα μιλήσει στο πάνελ μας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη συνεδρίαση εδώ, διότι και πέρσι είχε έρθει να μας εκθέσει τα μέτρα που ελήφθησαν για να καταπολεμηθεί η ενέργεια των νέων στην Ελλάδα. Ίσως επεκταθείτε αργότερα σε αυτά τα θέματα. Ο Ντανιέλ από την η ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση θα μας βοηθήσει ε, να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Πριν σας δώσω το λόγο, ε, αγαπητέ Πρόεδρε Κρεμαστινέ, ναι, θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, αν μου επιτρέπετε. Να θυμίσω ότι όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε να ε, ασχοληθεί με αυτό το θέμα τι συνέβη και πώς έγινε η όλη ε, διαδικασία. Ο πρόεδρος Φαν Ρόμπεϊ εκπονούσε τότε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την έκθεσή του, την ε, πρότασή του για το λεγόμενο οδικό χάρτη, επιμένοντας σε τέσσερις διαστάσεις που είχε εκείνο εντοπίσει για να προχωρήσουμε προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Δημοσιονομικά, θέματα χρηματοπιστωτικά, ε, δημοκρατίας και ένα τέταρτο που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά θα το θυμηθώ. Ε, θεωρήσαμε λοιπόν και εμείς ότι θα έπρεπε να επιμείνουμε να προσθεθεί και μια πέμπτη διάσταση που δεν είναι τίποτα το εξωγήινο ε, αλλά είναι πραγματικά η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Γι' αυτό σε μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις παραμονές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από ένα και πλέον έτος ε, συνεισφέραμε και εμείς στην κατάρτιση και εκπόνηση της θέσης του Κοινοβουλίου που πλέον ονομάζεται έκθεση Tyson και ζητούμε ρητά ε, να συμπεριληφθεί και να ληφθεί υπόψη και αυτή η πέμπτη διάσταση. Μετά από την πρωτοβουλία αυτή που υποστηρίχθηκε πάρα πολύ από τους κοινωνικούς εταίρους εκτός ε, των τυχών του Κοινοβουλίου, τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή ακριβώς να κάνει προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η ΔΕ Επιτροπή σε μια ανακοίνωσή της στα μέσα του περασμένου έτους ε, πρότεινε κάποια στοιχεία για την κοινωνική διάσταση. Γι' αυτό και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα ψήφισμα στην ανακοίνωση αυτή για να δώσουμε και τις δικές μας προτάσεις, το οποίο ψήφισμα γνώρισε πολύ μεγάλη υποστήριξη και υπερψηφίστηκε από 387 ε, υπέρ, 64 κατά και 58 αποχές. Εκεί θεωρούμε ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα πρώτο στάδιο, δηλαδή μια πρώτη φάση και μόνο για την υλοποίηση αυτής της πραγματικής ε, κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ. Ε, υπενθυμίζουμε βεβαίως την αρχή της επικουρικότητας που διέπει αυτά τα θέματα αλλά η κοινωνική δίτρα μας ε, ε, φάνηκε πάρα πολύ σημαντική για την εφαρμογή της, γιατί για μας τα κοινωνικά στοιχεία θα πρέπει να κυριαρχούν στην καρδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά σε όλες τις πρωτοβουλίες. Ε, χωρίς να υπενθυμίσουμε το άρθρο 9 ε, της Συνθήκης Λισαβόνας που δεν λαμβάνεται πολύ συχνά υπόψη. Θυμίζουμε ότι η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει ε, σε 26,6 εκατομμύρια. Είναι πολύ ανισχυτικό και 24,2% του πληθυσμού απειλείται με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ένωση. Άρα οι στόχοι για τη στρατηγική μας για το 2020 γνωρίζουμε ήδη από τώρα ότι δεν πρόκειται να εκπληρωθούν. Να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση. Θέλω να σε επιστήσω την προσοχή σε αυτό, διότι από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση πριν το τέλος τη θητεία τη τώρα να αναθεωρήσει ε, τη στρατηγική για το 2020 και ενδεχομένως να αμφισβητήσει την ίδια την ύπαρξη της πλατφόρμας για την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό δεν το θεωρούμε απλώς ανάρμοστο, αλλά και επί της ουσίας θεωρούμε ότι δεν είναι δουλειά τώρα της παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη λήξη της θητείας της να πάρει αποφάσεις που να καθοδηγήσουν τη στρατηγική για το 2020. Αν χρειαστεί κάτι τέτοιο είναι θέμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συζήτηση με το επόμενο κοινοβούλιο που θα εκλεγεί. Επανέρχομαι λοιπόν στη θέση του Κοινοβουλίου που αντέδρασε στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απορρίψαμε οποιαδήποτε εναρμόνιση ή ευθυγράμμιση προς τα κάτω ισοπαίδωση των κρατών μέλων ε, είναι ε, η περίφημη ρήτρα ε, της μη υπαναχώρησης. Τα γνωρίζουν αυτά οι η δική μας. Επίσης υπάρχει ένα θέμα δικτών για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ουσιώδης αυτή η πρόταση. αυτό θα ε, έρθει να συμπληρώσει τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα πρέπει να εξάγονται από την παρατήρηση για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατάρτιση της κοινή έκθεσης για την απασχόληση. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες αυτούς λοιπόν, θα πρέπει να βάλετε υπόψη και η διάσταση του φύλου και οι δείκτες να μετρούν και την ανεργία των νέων λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των 30 ετών, όπως συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο για την ε, εγγύηση για την νεολαία. Εκτός από τους πέντε δείκτες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς θα επιθυμούσαμε να προσθεθούν και άλλοι. Ξέρω ότι δεν θα πρέπει να το κάνουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο, να φορτώσουμε πάρα πολύ αυτό το ευχολόγιο, αλλά είναι και το θέμα της ένδυας των παιδιών, της πρόσβασης υπηρεσίες υγείας, καθώς επίσης και το ζήτημα του φαινομένου των αστέγων. Και ένα τέταρτο ακόμα το θέμα ε, της αξιοπρεπούς εργασίας. Και αυτά είναι δείκτες που θα πρέπει να ε, συμπεριληφθούν για να παρατηρούμε την κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση με την πιστότητα που χρειάζεται. Ζητούμε λοιπόν να συμπεριληφθούμε στην εκπόνηση αυτών των δικτών, αλλά κυρίως και επιμένω εδώ, η κοινωνική εταίροι στον κοινωνικό διάλογο θα πρέπει να συμμετέχουν ε, στον καθορισμό αυτών των στοιχείων. Επίσης θα θέλαμε το Συμβούλιο να ορίσει συγκεκριμένα ε, σημεία αναφοράς για δείκτες που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Κάτι που να αποτελεί ενός είδους προστατευτικό ε, ε, για την κοινωνική πρόνοια στην Ευρώπη. Επίσης καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνική διάσταση τη νομισματική ένωση και να υπάρχει η εθελοντική κινητικότητα των εργαζομένων. Κάποια στοιχεία συζητήθηκαν ήδη. Αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων και συνομιλιών μεταξύ μα. Ενδεχομένω να μην αντικατοπτρίζονται στα τελικά κείμενα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο, όμω εδώ μα απασχόλησαν τα στοιχεία αυτά. Συγκεκριμένα είναι δύο τα στοιχεία αυτά και είναι τα εξή αυτή τη στιγμή οριστούν αυτοί οι δείκτε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα στο πλαίσιο των ειδικών συστάσεων αναχώρα, οι οποίε συντάσσονται εκ των υστέρων και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε στη συζήτησή μα. Επίση, αρκετοί από εμά πιστεύουμε ότι δεδομένη τη αλληλεπίδραση τη οικονομική και κοινωνική διάσταση προ τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο μπορούσαν να υπάρχουν στοιχεία σταθεροποίησης αυτόματης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συγκεκριμένα περισσότερο στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες προτάσεις επιτάπητος, αλλά μία συγκεκριμένα αφορά τα μέλη των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης και αυτή μας αφορά, Δηλαδή το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας ε, για την κοινωνική προστασία με μια ελάχιστο επίδομα για την ανεργία οργανώσαμε στις 8 Ιουλίου του περασμένου έτους μία ακρόαση και σας προσκαλώ όλοι στο διαδίκτυο να κοιτάξετε τα στοιχεία της ακρόασης αυτής, ήταν ιδιαίτερα πλούσια και έθεσε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και μελλοντικά. Επίσης συζητήσαμε την προστεθέμενη αξία ενός τέτοιου μηχανισμού, στοιχεία που θα ξανασυζητήσουμε στις 12 και 13 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους στη συνεδρίασή μας. Αυτά λοιπόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όταν κάποτε ο όπως όταν κάποτε ο κύριος Ντελόρ είχε ζητήσει τη συμβουλή αυτής της Επιτροπής, θα ζητήσουμε και εμείς λοιπόν από την ΕΟΚΕ να μας δώσει τη συνεισφορά της για τη λειτουργία για τη λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου. Όχι τι λεπτομέρειε του κοινωνικού διαλόγου, αλλά πώ θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τον κοινωνικό διάλογο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εδώ και μέρε ακούμε ότι χρειάζεται κοινωνικό διάλογο, τον χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά επειδή δεν βλέπουμε κάτι χειροπιαστό, εμεί θέλουμε με αυτή την πρωτοβουλία να καταλήξουμε και σε νέε προτάσει. Σα ευχαριστώ, με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά όπω θα γνωρίζετε πολλοί από εσά, πρόκειται για ένα θέμα που πραγματικά μα απασχολεί ιδιαιτέρω θα ήθελα για αυτό το λόγο η συζήτηση με τα εθνικά κοινοβούλια να επικεντρώνεται στην ουσία. Δεδομένων όσων είπα και από την αρχή για την κατανομή αρμοδιοτήτων. Με μεγάλη χαρά τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κρεμαστινό ώστε ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής να μας ε, παρουσιάσει τις δικές του απόψεις. Έχετε πέντε λεπτά, πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Περές. Είμαι ε, ε, μεγάλη χαρά προεδρεύω μαζί με την κυρία Περβάς Περές σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνεδρίαση και τόσο ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την ανεργία και τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Και φυσικά έχω δίπλα μου τον Υπουργό Εργασία ε, της Ελλάδας, τον ε, φίλο τον κύριο Βρούτση, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια τεράστια προσπάθεια στην κατεξοχή χώρα που πλήττεται από την ανεργία ε, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη κρίση. Και θα είμαι θα ευτυχής να ακούσουμε τις προσπάθειες αυτές που καταβάλει. Όμως θα πρέπει να πω ότι και πέρσι σε αυτή την αίθουσα ακούστηκαν περίπου τα ίδια λόγια ότι για τις χώρες του Νότου και ειδικότερα για την Ελλάδα ε, τις χώρες του Νότου που πλήττονται από την ενεργία ε, λέχθηκε τότε ένας στους τρεις Έλληνες ζει κάτω από το όριο της στόχιας η ανεργία έχει ξεπεράσει τότε το 26% τώρα βρίσκεται στο 27% με ένα από τους δύο νέους να βρίσκεται στο εργασιακό περιθώριο μια στις δύο οικογένειες πέρσι αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι της. Ε, μία στις δύο οικογένειες πέραν το ότι αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι της φορολογείται και περισσότερο. Η φορολογία κατά ανάγκη να αυξάνεται. Οι μισθοί μειώνονται, οι τιμές παραμένουν ψηλές στα κατανοητικά αγαθά. Ε, όμως ε, μοιάζει όλη η ιστορία να οδηγεί σε διέξοδο και όλοι ε, επαναλαμβάνουν τη μαγική λέξη που λέγεται ανάπτυξη. Όταν υπάρξει ανάπτυξη τότε όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν και βεβαίως και η ανεργία θα ελαττωθεί, θα μειωθεί, θα εξαφανιστεί. Όμως, ε, όμως τι είδου ανάπτυξη προτείνεται για τις χώρες του Νότου. Sorry. Δεν υπάρχει μετάφραση. Δεν υπάρχει. There ε, Υπάρχει άλλο μικρόφωνο. Αναμένω, υπάρχει και άλλο μικρόφωνο αναμένο, γι' αυτό δεν ακούγεται καλά κύριε Κρομαστινή. Okay. Can we have a test with the German... Είναι γερμανική καμπίνα, μπορείτε να το ελέγξετε κύριε Τόμασμάν αν είναι εντάξει, παρακαλώ. Όχι, ε, δεν γίνεται αυτό. Είναι ανοιχτά δύο μικρόφωνα είναι και άλλο μικρόφωνο ανοιχτό στην αίθουσα. Ici, je vois pas l'autre Πρόεδρος, δεν βλέπω άλλο μικρόφωνο αναμένο. Ποιος έχει αναμένο μικρόφωνο. Παρακαλώ να το ασβήσετε, μόνο ο μιλητής να ακούγεται. Α ε, Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Ε, και πάλι θα επαναλάβω τα ίδια. Ε, δεν ξέρω. It's okay. It's okay. Ε, από... <laughs> από ποιο σημείο δεν έχετε ακούσει. Από την αρχή ή από τώρα. από τώρα. Ε, θα επαναλάβω λοιπόν τα ίδια κατά ανάγκη. Ε, είπα ότι και πέρσι σε αυτή την αίθουσα είχαν ακουστεί περίπου τα εξή πράγματα για τις χώρες του Νότου και ειδικότερα για την Ελλάδα. Ότι ένας στους τρει Έλληνες ζει κάτω από το όριο τη στόχιας. Ότι οι άστεγοι και τα συσίτια πολλαπλασιάζονται. Η ανεργία για πέρσι είχε ξεπεράσει το 26% και είναι γύρω στο 27% με ένα στους δύο νέους να βρίσκονται στο εργασιακό περιθώριο, να είναι άνεργοι. Μια στις δύο οικογένειες να αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι της. Παράλληλα η φορολογία να αυξάνεται, οι μισθοί να μειώνονται και οι τιμές να παραμένουν ψηλές στα καταναλωτικά αγαθά. Και όλοι επαναλαμβάνουν ότι η μαγική λέξη, τη μαγική λέξη ανάπτυξη και όταν υπάρξει ανάπτυξη τότε όλα αυτά τα δεινά θα εξαφανιστούν και η ανεργία θα αντιμετωπιστεί, θα εξαφανιστεί και η φορολογία θα πέσει και οι τιμές θα γίνουν ορθολογικές. Όμως τι είδου ανάπτυξη. Το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί ουσιαστικά να επιχορηγήσει τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες για να υπάρξει ανάπτυξη. Δεδομένου ότι ε, οι τράπεζες του Νότου βρίσκονται σε αδυναμία να χρηματοδοτήσουν με δάνεια τις επιχειρήσεις και ειδικότερα οι τράπεζες της Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η ανάπτυξη η τριτοκοσμικού τύπου. Δηλαδή όταν όλοι, όταν τα πάντα μηδενιστούν, όταν δεν υπάρχει ζωή, τότε κάποιοι θα διαφερθούν για να επενδύσουν στη χώρα αυτή. Αλλά αυτή δεν θα είναι μια χώρα της Ευρώπης ή δεν θα είναι οι χώρε της Ευρώπης του Νότου, θα είναι οι χώρε της Ευρώπης του τρίτου κόσμου. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα να αποτελεί θέμα συζήτησης. Ε, βεβαίως ε, υπάρχει και μία άλλη ανάπτυξη. Αυτή την οποία ξέρει και έχει επιχειρήσει η Ευρώπη σε άλλες περιόδους. Παραδείγματος χάρη ε, ακούστηκε στην προεκλογική περίοδο στη Γερμανία από το s που τώρα αυτή τη στιγμή συγκυβερνά ότι για τις χώρες του Νότου και ειδικότερα την Ελλάδα θα πρέπει να επαναληφθεί ε, το σχέδιο Marshall κατά αναλογία που είχε υπάρξει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν η Γερμανία ήταν ισοπεδωμένη και η οποία χρηματοδοτήθηκε για να αναπτύξει τη βιομηχανία της και να ξεπληρώσει κατά κάποιο τρόπο τα δάνειά της όταν η βιομηχανία θα απέδιδε καρπούς. Αυτή η ανάπτυξη είναι ενδεδειγμένη για τις χώρες του Νότου και ειδικότερα για την Ελλάδα. Και λέω την Ελλάδα όχι διότι και εγώ είμαι Έλληνας και ο Υπουργός είναι Έλληνας, αλλά είναι η κατεξοχήν πληττόμενη χώρα. Μπορεί παραδείγματο χάρη με τέτοιου είδου ανάπτυξη να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί ο τουρισμό, διότι η χώρα στερείται υποδομών. Εάν δηλαδή με την ανάπτυξη δημιουργηθούν μαρίνε ή λιμάνια, τότε τα ελιμενιζόμενα πλοία θα τριπλασιαστούν και θα αυξηθούν, τότε τα γιότ θα πολλαπλασιαστούν και τότε η Ελλάδα που έχει αποδεδειγμένα το καλύτερο κλίμα και τις καλύτερες θάλασσες θα είναι θεωρητικά από τις πρώτες χώρες της τουριστικής Ευρώπης, που σήμερα δεν είναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλο, αν θέλετε, επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν εκδηλώνεται. Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί και για άλλους τομείς, όπως είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, όπως είναι ο υποθαλάσσιος πλούτος, όπως είναι η αιωλική ενέργεια, διότι στην Ελλάδα φυσάνε κάθε μέρα άνεμοι πάνω από 7 μποφόρ, ε, στο Αιγαίο κατεξοχήν, στο Αιγαίο Πέλαγος και κατά συνέπεια θα μπορούσε να είναι αυτάρκης ακόμα και ενεργειακά. Άρα λοιπόν η, αυτού του είδους η προσπάθεια θα ήταν μια προσπάθεια που θα μπορούσε να αποδώσει ουσιαστικά και μέσα στα προσεχή χρόνια. Ε, όμως ε, εγώ ε, έκανα απλώς ορισμένες νήξεις συμπροεδρεύοντας με την κυρία Περές και δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό Εργασίας της Ελλάδας, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος ε, θα σας περιγράψει το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ, κύριε Κρεμαστίνα. Για την ελληνική προεδρία λοιπόν θα σας δώσω το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ελπίζουμε το μήνυμα που θα μας αποστείλετε είναι ως ε, υπεύθυνος της προεδρεύουσας χώρας να μας πείτε για την κοινωνική διάσταση της ε, Νομισματικής Ένωσης η οποία ελπίζουμε ότι είναι κάτι που θα καλύψετε κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. Ένα εξάμενο ιδιαίτερο ε, δεδομένων των συμπερασμάτων του Συμβουλίου από τον περασμένο Δεκέμβριο ή Επίσης και της προοπτικής των ευρωεκλογών αυτή την άνοιξη. Δεν θέλουμε να παραμεληθεί το θέμα αυτό και πραγματικά θα θέλαμε να ακούσουμε πώς θα το καλύψετε εσείς κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας σας, που είναι γεμάτη προκλήσεις. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Μπερές, Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Επιτροπής για την Απασχόληση, κύριε Κρεμαστινέ, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, εκ προημίου θέλω να δηλώσω ενώπιόν σας ότι αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τη χώρα μου την Ελλάδα με την ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αλλά και ταυτόχρονα έχοντας πλέον τη νέα ιδιότητα του Υπουργού που στον κρίσιμο αυτό τομέα θα έχει την ευθύνη λόγω της προεδρίας, της ελληνικής προεδρίας να κρατήσει το τιμόνι στα κρίσιμα αυτά ζητήματα για το επόμενο εξάμεινο. Απευθύνομαι λοιπόν σε εσά που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είστε η πιο κρίσιμη ομάδα μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα, στο θεσμικό ευρωπαϊκό σύστημα που διαμορφώνεται ως κλειδί το διάλογο στην Ευρώπη. Από εδώ περνάνε πολύ κρίσιμα και σημαντικά ζητήματα. Και απευθύνομαι και σε εσά που την τρέχουσα θητεία, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι τι ευρωεκλογέ, έχετε πραγματικά επιδείξει ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο αφήνει έντονο το θετικό αποτύπωμά του παρά την αρνητική συγκυρία που έτρεξε αυτή την περίοδο της κρίσης. Επιπλέον, απευθυνόμενος και προς την κυρία Πρόεδρο στα ερωτήματα που έθεσε, θέλω να σας πω ότι παρά την κρίσιμότητα των στιγμών η ελληνική προεδρία θα είναι μια πολύ καλή προεδρία. Και θα κάνουμε, κυρία Πρόεδρε, ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι και τα κοινά οραματά μας μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Η ελληνική προεδρία θα είναι μια καλή προεδρία. Και ελπίζουμε με τη βοήθεια όλων και τη συνδρομή όλων οι κοινοί στόχοι που έχουμε θέσει να ευοδοθούν στο τέλος αυτής της προεδρίας. Ξέρουμε ότι πολλά πράγματα είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν εκκρεμότητες δηλαδή που έρχονται από το παρελθόν, όμως αυτά τα ζητήματα θα τα παραδώσουμε στην επόμενη Προεδρία, στην Ιταλία, έχοντας κάνει σημαντικά βήματα. Και ελπίζουμε ότι πολλά άλλα ζητήματα που έχετε θέσει και κληρονομούμε από το παρελθόν θα τα επιλύσουμε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο ρόλος αυτός, δηλαδή της Επιτροπής, αποκτά κρίσιμη σημασία. Γιατί σήμερα η Ευρώπη πραγματικά βιώνει μια πολύ σημαντική ή πολλές σημαντικές προκλήσεις, πρωτόγνωρες θα έλεγα. Η κρίση έχει θέσει ενώπιόν μας μια σειρά αποζητήματα που ζητούν άμεση, αποφασιστική και αποτελεσματική δράση. Και το καταλαβαίνουμε όλοι. Πέντε χρόνια τώρα αποκάλυψαν ότι η οικονομική πορεία που ακολουθούσε η Ευρώπη παρουσίαζε ρογμές. Μάλιστα η πορεία αυτή δεν διασφάλιζε τη βιωσιμότητα ούτε της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ούτε του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η κρίση ανέδειξε διαρθρωτικές αδυναμίες σε διάφορα επίπεδα της Ένωσης που ζητούν τώρα την άμεση ανταπόκρισή μας, τώρα που εμφανίστηκαν μπροστά μας. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει ήδη το πέμπτο έτος της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μια στρατηγική για την έξυπνη, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη που προάγει την ένταξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Η συγκεκριμένη στρατηγική συνιστά ένα κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στοχεύει αφενός την καταπολέμηση των αδυναμιών του ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου και αφετέρου στη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθήκων για την επίτευξη των στόχων της. Σήμερα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταδεικνύουν ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξαν ενθαρρυντικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης. Μετά τη συρρήκνωση της οικονομίας, μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2013, η ευρωπαϊκή οικονομία επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά το δεύτερο τρίμηνο. Το πραγματικό ΕΠ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο εμφανίζεται μπροστά μας. Η ανάκαμψη αυτή βέβαια δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι εξακολουθεί να είναι επισφαλής και δεν αφορά στον ίδιο βαθμό όλα τα κράτη-μέλη. Επιπλέον είναι ακόμα ιδιαίτερα πρόωρο να διαπιστώσουμε με βεβαιότητα ότι συμπέρασμα ότι αυτή θα είναι σταθερή και θα διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική κατάσταση της Ευρώπης αρχίζει για πρώτη φορά να δείχνει θετικά σημάδια. Επιτρέψτε μου εδώ, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και όχι άδικα, να κάνω κάποιες επισημάνσεις για τη χώρα μου την Ελλάδα. Στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη εμφανίζονται και εκεί τα αντίστοιχα πρώτα θετικά σημάδια. Η ανεργία για παράδειγμα που παρότι έχουμε το δυσμενές προνόμιο να έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, εμφανίζει μέσα στο 2013 εμφάνισε σταθερής, σταθερές τάσεις σταθεροποίησης. Κατά την επόμενη περίοδο εκτιμούμε και το λένε και οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και δικά μας εργαλεία που έχουμε ότι θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία αποκλιμάκωσης μέσα στο 2014 της ανεργίας. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ορθής εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που κάναμε με συνέπεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια όπως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι και στη χώρα μου μπορούμε να πούμε ότι η δημοσιονομική εξυγένση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν θέτουν συνολικά τα θεμέλια της ανάκαμψης. Και εμείς στην Ελλάδα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της παρατεταμένης ύφεσης, ξεκινήσαμε ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών Στη διεθνή κατάταξη του ΟΣΑ, παραδείγματο χάρη, η Ελλάδα κατατάσσεται ήδη στην πρώτη θέση όσο αφορά την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών. Και τα αποτελέσματα φάνηκαν. Σύμφωνα με όλες τις έρευνες, ανακτήσαμε ήδη τη χαμένη μας ανταγωνιστικότητα. Από το 2002, ενώ μηδενίσαμε το έλλειμμά μας στο εμπορικό ισοζύγιο. Ενώ επιπλέον κάτι πολύ σημαντικό, μετά από 10 χρόνια εμφανίζουμε για πρώτη φορά πρωτογενές πλεόνασμα. Κάτι το οποίο φαινόταν αδύνατον και πολλοί στοιχημάτιζαν ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών. Ωστόσο εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι φιλικές στην ανάπτυξη, να έχουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική μας, η στρατηγική της Ευρώπης 2020 και πάνω απ' όλα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την κύρια πρόκληση που θέτει πραγματικότητα. Δηλαδή να συνδυάζουν την κοινή προσπάθεια για δημοσιονομική σταθερότητα με πολιτικές για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Αυτό γιατί όσο θετικές και αν είναι οι εξελίξεις, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρουσιάζουν κατά κανόνα υστέρηση σε σχέση με τις εξελίξεις στο ΑΕΠ. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να οδηγήσει μόνο σταδιακά σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Φέτος η ανεργία παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες και η απασχόληση εξακολούθησε να μειώνεται. Ωστόσο κατά τους τελευταίους μήνες οι συνθήκες στην αγορά εργασίας άρχισε, άρχισαν να σταθεροποιούνται. Έως το 2015 προβλέπεται συγκρατημένη μείωση της ανεργίας περίπου στο 10,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 11,8% στην Ευρωζώνη. Ωστόσο όμως, εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Συνεπώς, στον τομέα αυτό χρειάζεται οραματισμός και αποφασιστικότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί. Πολιτικών που στο επίκεντρό τους έχουν την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη περίοδο, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Είναι η χρονιά των ευρωεκλογών, της τοποθέτησης της νέας Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014 και της τοποθέτησης και του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παράλληλα, κρίσιμες εξελίξεις έχουμε και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Το κόστος από την καθυστέρηση υλοποίησης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και δράσεων έχει υπάρξει ενίοτε αρκετά υψηλό. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας έχουν ως συνέπεια την όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων, την υπονόμευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ένωσης, τον περιορισμό των εισοδημάτων και της ενεργού ζήτησης. Επιπλέον, δρούν ανασταλτικά αναφορικά με την παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό μας. Αδυνατίζουν την πολιτική υποστήριξη προς τις αναγκαίες δράσεις για το ξεπέρασμα της κρίσης, ενώ ενισχύουν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων, όπως πριν από λίγο σας περιέγραψε και ο πρόεδρος ο κύριος Κρεμαστινός. Σε μια τέτοια συγκυρία είναι ακόμα πιο επίγουσα η εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ακριβώς τώρα είναι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη συνθήκη όπως και τους στόχους της Ευρώπης 2020. Όχι μόνο επειδή αυτό είναι το παγκόσμιο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, αλλά κυρίως επειδή αυτή είναι η καρδιά του κοινωνικού συμβολέου που διασφαλίζει την πολιτική μας σταθερότητα και την κοινή μας πορεία στο μέλλον. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο μέσα από τη συλλογική μας δράση μέσα από ένα βέλτιστο συντονισμό μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Να διασφαλίσουμε ότι η απασχόληση και οι προκλήσεις στο κοινωνικό τομέα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και άμεσα. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο οι αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Όπως γνωρίζετε, το σύνολο των ευρωπαϊκών οργάνων αναγνωρίζει την κρισιμότητα της εμβάθυνσης της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ η βελτίωση της παρακολούθησης των εξελίξεων στην απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα είναι επίγουσα, είναι αναγκαία. Γιατί έτσι μπορούμε να διακρίνουμε έγκαιρα τις απειλές και τις κοινωνικές ανισορροπίες όπου αναδύονται, έτσι ώστε να αντιδρούμε, να λειτουργούμε άμεσα. Ήδη στον τομέα της Νομισματικής Ένωσης έχουν διαμορφωθεί μια σειρά από εργαλεία τα οποία προσφέρουν τις δυνατότητες για πραγματικές, γρήγορες και αποτελεσματικές προσαρμογές. Με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τις αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, φιλοδοξούμε ότι θα διαμορφώσουμε παρόμοιες διαδικασίες και στον κοινωνικό τομέα. Ασφαλώς, η ορθή και έγκαιρη παρακολούθηση των εξελίξεων αποτελεί ένα μέρος της ιστορίας, διότι σημασία για την ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης έχει η διαμόρφωση διαδικασιών που θα επιτρέπουν την έγκαιρη πρόβλεψη και την αποτροπή εξελίξεων που οδηγούν σε ανισότητες και δυσλειτουργίες. Εξελίξεις που σε τελική ανάλυση αποτελούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του συνόλου της ΟΝΕ, την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Μετά το τελευταίο έψκο του Δεκεμβρίου ενσωματώθηκε, και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, στο τρέχον ευρωπαϊκό εξάμεινο ο πίνακας αποτελεσμάτων δικτών απασχόληση και κοινωνικών δικτών scoreboard. Στόχος της ελληνικής προεδρίας. Και κυρία Πρόεδρε πιστέψτε με θέλουμε να το κάνουμε πράξη. It's the time, eh? about minutes. finished. Mm. Είναι, είναι σε συνεργασία με όλους σας να ολοκληρώσουμε αυτή την πρόκληση και την προτεραιότητα. Σε αυτά που είπε η κυρία Μπέρες, δηλαδή το να προσθέσουμε επιπλέον κοινωνικούς δίκτες συμφωνώ. Όπως επίσης είχα πει και στο ΕΠΣΚΟ ότι υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοδείκτες όπως ο δείκτης που έχει να κάνει με τη δημογραφία σε μια Ευρώπη που γερνάει, το δημογραφικό πρόβλημα. Όλα αυτά είναι προκλήσεις ανεκτές, στις οποίες θέλω να διαβεβαιώσω άλλη μία φορά την Επιτροπή ότι αυτά και μαζί με τις άλλες προτεραιότητες θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα ενελοποιήσουμε και να τα κάνουμε πράξη στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, για την επισκόπηση αυτή και την περιγραφή της ε, κατάστασης και στην Ελλάδα αλλά και για την Προεδρία για αυτό το θέμα της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ και πώς θα ληφθεί υπόψη. Τώρα, ε, από πλευράς Εθνικών Κοινοβούλων. Ζητήσαμε από την κυρία Ντανιέλου Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης που έχει κάνει ε, μεγάλο έργο για αυτά τα θέματα να έρθει εδώ να μας ε, καταθέσει τη μαρτυρία της και να συνεισφέρει στη συζήτηση που θα ανοίξει ε, από τα κοινοβούλια μας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι εδώ σήμερα. Νομίζω οι διακοινοβουλευτικέ συνδυάσει είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μπορέσουμε να έχουμε μια εύστοχη ανταλλαγή απόψεων και να μπορέσουμε να θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Κάποια σημεία αναπτύχθηκαν ήδη από του προηγούμενου αγορητέ, όμω επιτρέψτε να τα θίξω κι εγώ. Γιατί να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση τη Νομισματική και Οικονομική Ένωση, ε, την παραμονή των ευρωεκλογών. Νομίζω δεν χρειάζεται καν να το θέσουμε το ερώτημα. Είναι αυτονόητο. Από το 2008 βλέπουμε ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει του μηχανισμού συντονισμού τη μακροοικονομική ε, σύγκληση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού αλλά τι μπορούν να καταλάβουν οι πολίτε μα από όλα αυτά που κάνουμε. Μόνον ότι συνεχίζουν να υποφέρουν και δεν βρίσκουν δουλειά. Από αυτήν λοιπόν την άποψη, το να ορίσουμε ένα σύνολο πρωτοβουλειών που θα ενισχύσουν την κοινωνική διάσταση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ο μόνο τρόπο νομίζω για να είμαστε κατανοητοί, ε, να αντιληφθούν οι πολίτε μα τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε του αριθμού στα χέρια μα. Ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού απολύεται από τη φτώχεια, συμπεριλαμβανομένης τη Γερμανία. Ο πληθυσμό που είναι φτωχός στη Γερμανία, οι φτωχοί εργαζόμενοι είναι πολλοί. Ε, να μην επανέλθω σε πράγματα που υπόθηκαν χθε στην Ολομέλεια, αλλά ένα στου πέντε νέου δεν έχει δουλειά σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μαζί με, φυσικά με κάποιε πιο ακραίε εκδηλώσει στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ε, η χώρες που βρίσκονται επισήμως σε πρόγραμμα προσαρμογής η Ισπανία και η Πορτογαλία ε, γνωρίζουν αυξημένες συνθήκες φτώχειας. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα πάνε καλύτερα στους οικονομικούς δείκτες ότι ο πληθυσμός είναι καλύτερα. Ε, κάθε πολιτική λοιπόν που δεν αντισταθμίζει τι συνέπειε τη κρίση είναι πολιτική εθνική λιτότητας. Ξέρουμε ότι κάποια μέτρα έχουν επιβληθεί από την Τρόικα πολύ απότομα. Το ίδιο το Νομισματικό Ταμείο το παραδέχεται. Εάν δεν υπάρχει θελοντική δράση υπέρ τη απασχόληση και τη κοινωνική επένδυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι και οπουδήποτε χρειαστεί να εκλεγούμε. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την κοινωνική Ευρώπη. Αυτό είναι η πρώτη ε, ανάγκη, η πρώτη προτεραιότητα για να έχει νόημα αυτή η συλλογική και δυσχερή οικοδόμηση. Θα πρέπει να πείσουμε του πολίτε μα ότι εργαζόμαστε προ όφελό του και σε αυτόν τον τομέα για στη δική τους υπηρεσία και όχι μόνο στην υπηρεσία των χρηματοπιστωτικών αγορών και των εγωισμών τους. Όπως είχε πει ο Επίτροπος Άντορ, όπως και εσεί ίδια κυρία Πρόεδρε, πρέπει να δώσουμε μια σημαντική όθηση, αποφασιστική όθηση προς αυτή τη νέα κατεύθυνση. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται βεβαίω και σε τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου του 2013 είχε τονίσει την ανάγκη να ενισχύσουμε το συντονισμό, την ε, εποπτεία των κοινωνικών ε, πολιτικών στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση σε αυτό το τομέα. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να αντιμετωπίσει τις ε, δυσκολίες που προκαλεί η οικονομική προσαρμογή για κοινωνικές διαστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη εποπτεία των πολιτικών και των κοινωνικών του συνεπειών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε διδάγματα από την αλληλεγγύη που επιβάλλει η ε, ο συντονισμό επίπεδο ευρωπαϊκού προπολογισμού και να συνδυάσουμε τα εθνικά, τις εθνικές προσπάθειες για την ε, κοινωνική πολιτική στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο συγκεκριμένο εντοπισμός των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων και απασχόλησης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κάτι που ήδη έχουμε ε, θέσει ως προτεραιότητα με τη δημιουργία πέντε νέων δικτών για να δούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της μακροοικονομικής προσαρμογής. Η Επιτροπή τον απολογισμό που πρότεινε με τον μηχανισμό αγιοσφαιρετοποίηση είναι να δούμε την κατάσταση τη απασχόληση και των κοινωνικών συνθήκων στι χώρε που έχουν πληγεί. Ακόμη και με μηχανισμού κοινωνική προσαρμογή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε να προωθηθούν οι πρακτικέ αριστεία σε διάφορα κράτη-μέλη. Όταν βλέπουμε στην Ελλάδα, όπω το υπογράμμισε και ο Υπουργό, ένα μεγάλο μέρο των Ελλήνων που δεν έχουν πρόσβαση σε καμία ε, μορφή κοινωνική πρόνοια, θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει. Όχι μόνο οι Έλληνε, Έχουμε λοιπόν νομίζω ε, κάνει ένα βήμα ακόμη. Τον περασμένο Νοέμβριο το Κοινοβούλιο δυστυχώς ενέκρινε ένα ψήφισμα λιγότερο φιλόδοξο από αυτό που αρχικά προτινόταν από την Επιτροπή. Και εσείς Πρόεδρε, δικαίω αγωνιστήκατε για να είστε δυνατόν φιλοδοξότερο το ψήφισμα αυτό. Λέγατε ότι χρειάζεται νέα εξισορροπή μεταξύ των οικονομικών και, πολιτικών και κοινωνικών πολιτικών, προκειμένου να υπάρξει σύγκληση όχι μόνο υπό την ε, σκοπιά των μακροοικονομικών όρων, αλλά και των κοινωνικών. Χωρί αυτό, το μέλλον τη Ευρωζώνη δεν θα είναι ε, μακρό και ομαλό. Αυτό νομίζω το συμμερίζονται και οι επιτροπέ Κοινωνικών Υποθέσεων. Δυστυχώς αποδυναμώθηκε το ψήφισμα. Ε, δεν αναφέρεται πλέον στα μέτρα λιτότητας. Διαγράφηκε ένα εδάφιο που λέει ότι η υποτίμηση νομισμάτων για σκοπούς εξισορρόπησης μακροοικονομικής δεν λαμβάνει υπόψη την ελεξάρτηση μεταξύ των κρατών και τις κοινωνικές συνέπειες. Το ίδιο με το πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είναι ικανοποιητικό στο σύνολο δικτών που έχει επιλέξει. Επίσης, ε, ο κοινωνικός πυλώνας δεν αναφέρεται, ενώ το Συμβούλιο το Δεκέμβριο είχε ζητήσει να ενσωματωθεί στην ΟΝΕ. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ένα αρνητικότατο μήνυμα προς τους πολίτες μας. Όμως, Παρόλα αυτά, και θα πρέπει να δούμε τα θετικά, το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε επιπλέον δείκτες στον πίνακα αποτελεσμάτων. Κοινωνικούς δείκτες. Αυτό νομίζω δικαίως ζητήθηκε και άρχισε ήδη να εφαρμόζεται σε επίπεδο γαλλικού κράτους. Η φτώχεια των παιδιών, η πρόσβαση στην κοινωνική, προ... στις, ε, στην οικονομική περίθαλψη, η... το φαινόμενο των αστέγων, η αξιοπρεπής εργασία, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με αποσπασμένου εργαζομένους που εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες, Όλα αυτά είναι λογικά πράγματα που ζητούνται για την κοινωνική προστασία στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί σας στηρίζουμε, κυρία Μπερές. Και εγώ και η συνάδελφος υπεύθυνη για τα θέματα αυτά στην ε, ε, Γαλλική Βουλή, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, είμαστε στο πλευρό σας. Στις 8 Φεβρουαρίου άλλωστε θα έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο κειμένου για τα θέματα αυτά. Ελπίζω ότι οι παρόντες ευρωβουλευτές θα, θα μπορέσουν να έχουν μια πλούσια συζήτηση μαζί μας. Θα θέλαμε λοιπόν να τονιστεί η κοινωνική διάσταση αυτού του εξαμήνου, του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Θα πρέπει να είναι παρούσα καθ' τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι μόνο να εξετάζεται μια φορά χρόνο μαζί με την αύξηση. Ο πίνακα αποτελεσμάτων για την κοινωνική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να είναι ένα σύνολο από διαπιστώσει, αλλά να είναι ένα εργαλείο για να ορίσουμε προσανατολισμό για τι οικονομικέ μα πολιτικέ με κοινωνική τροχιά. Θα πρέπει οι χώρε να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική πτυχή των οικονομικών του πολιτικών, να λαμβάνουν υπόψη την ποιότητα τη απασχόληση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στη διαβιωμάτιση, καθώ και την καταπολέμηση τη φτώχεια. Σε ό,τι αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινωνικοί δείκτε πρέπει να συμπληρωθούν. Δεν θα επανέλθω στην εξαιρετική έκθεση του κ. Γκουτιέρε Πιέτο, ο οποίος ε, μιλά για δείκτε που αφορούν τη φτώχεια των παιδιών, για τον δείκτη τη εξωπροπού εργασία και τη κάλυψη των ζωτικών αναγκών, αλλά θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και τον συντελεστή της ε, τον συντελεστή των ανισοτήτων ε, για τα εισοδήματα. Θα πρέπει οι κοινωνικοί δείκτες να αποκτήσουν επίσης δεσμευτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε την εποπτεία των ε, μακροοικονομικών και οικονομικών ελλημάτων με την παρατήρηση των κοινωνικών ανισορροπιών επίσης. Οι κοινωνικές υποθέσεις και η απασχόληση θα πρέπει να είναι αντικείμενο ε, πολυμερούς παρακολούθησης ώστε να μπορέσουν να διαδοθούν και οι καλύτερες πρακτικές. Επίσης, μια δεύτερη ιδέα σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση για την κοινωνική διάσταση τη ΩΝΕ. Επειδή υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών τη Ευρωζώνη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα στην διακυβέρνηση τη ΩΝΕ. Ε, για το σκοπό αυτό, η δυνατότητα που θα δοθεί στον, ε, στη Σύνοδο της, ε, των Υπουργών της Ευρωζώνης θα είναι να ασχοληθούν όχι μόνο με οικονομικά θέματα, αλλά να προβλέψουν και την ε, τακτική ε, σύνοδο των Υπουργών που ασχολούνται με κοινωνικές υποθέσεις και την απασχόληση. Για την ώρα αυτό δεν έχει γίνει. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει ό,τι μπορεί. Ε, η διάσκεψη που προβλέπεται στο άρθρο 13 είναι ένα πρωτοβήμα, ώστε να υπάρξει ένα πρώτο διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίων για τα θέματα αυτά αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα κανόνα πιο σαφή, ώστε τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα και ένα χρονοδιάγραμμα. Και μια τρίτη ιδέα. Νομίζω θα πρέπει χωρί κανένα δισταγμό να προβλέψουμε ένα σύστημα σταθεροποίηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σύστημα που να, να προβλέπει ένα επίδομα ανεργία και έναν ελάχιστο κατώτατο μισθό. Αυτό το περιμέναμε πολύ. Στη Γαλλία έχουμε τον κατώτατο μισθό, τον λεγόμενο ΣΜΙΚ. Η Γερμανία προβλέπει κάτι τώρα για το μέλλον, αλλά Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια τέτοια αναφορά, ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν κατώτατο μισθό, νομίζω ότι αυτό θα έδινε ελπίδα σε όλους μας τους πολίτες. Διότι ο κατώτατος μισθός, ακόμα και αν σε διάφορες χώρες υπολογίζεται διαφορετικά, θα έδινε μεγάλη ελπίδα στους ε, πολίτες είναι σημαντικό για τη Ρουμανία, ακόμη και αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό το ποσό στην Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία. Έτσι λοιπόν ξέρουν οι άνθρωποι, θα ξέραν οι άνθρωποι ότι δεν θα βυθιστούν στη φτώχεια, ακόμη και αν χάσουν τελείω τη δουλειά τους. Ε, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τα πρότυπα του παρελθόντος. Νομίζω η κυρία Μπερέση έκανε πολύ ακριβείς προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θα πρέπει την παραμονή των ευρωεκλογών να κινητοποιηθούμε όλοι, να αξιοποιήσουμε όλα μας τα μέσα ώστε να μπορέσουμε να ε, προωθήσουμε αυτή την κοινωνική Ευρώπη. Κάτι που έχει γίνει μια απαραίτητη πλέον διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο σας και ε, Υπήρξε κάποια σύγχυση ε, ε, ως προς την έναρξη της συνεδρίασης, τι ώρα αρχίζαμε δηλαδή και δεν ακούσατε την αρχική μου παρέμβαση που συνέπεσε σε μεγάλο βαθμό με τα όσα είπατε εσείς. Σε ό,τι αφορά το κατώτατο ή ελάχιστο εισόδημα, εδώ στο Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών μας ε, προσπαθούμε και φροντίζουμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε μισθό και εισόδημα διότι ε, είναι άλλη τάξεως ε, ζητήματα κάθε φορά αυτά. Τίθετε πάντως το θέμα και συζητείτε. Έχετε ζητήσει το λόγο πάρα πολύ ήδη με ε, τα κίτρινα χαρτιά αυτά. Παρακαλώ όποιος θέλει να μιλήσει σε αυτό το θέμα για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ να ζητήσει το λόγο. Θα είμαι φρικτή πρόεδρος, δηλαδή θα έχετε ένα δίλεπτο μόνο να μιλήσετε. Είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουν όλοι το λόγο και να εκφραστούν. Και να μπορέσουν να συνεισφέρουν σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Θα δώσω μέσω το λόγο σε εκείνον που θα δώσει και το καλό παράδειγμα, ε, Dominic Hannigan από την Ιρλανδική Βουλή. Παρακαλώ. vous avez minutes λεπτά έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ιρλανδία επικροτεί την πρόταση της Κομισιόν να συμπεριληφθεί κοινωνική διάσταση στην ΟΝΕ και στην δημοσίευση του σχεδίου των κοινωνικών δικτών. Και κυρία Πρόεδρε, πιστεύουμε ότι μπορούν να συμπεριληφθούν κάποιοι επιπλέον δείκτες. Η Επιτροπή μου τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο είχαν μια σειρά συνεδριάσεων για να συζητηθούν οι προτάσεις της Κομισιόν και καλέσαμε μέλη ε, των ε, ε, οργανώσεων απασχόλησης του Συμβουλίου Γυναικών και τους ρωτήσαμε τι πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες. Αναγνώρισαν ότι θα πρέπει να υπάρχει περιορισμένος αριθμός δικτών. Θέλουμε όμως να περιλαμβάνονται θέματα ισότητας, ιδιαίτερα την διαφορά ανάμεσα στους μισθούς ανδρών και γυναικών και επίσης ε, δείκτες που να αφορούν τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, επίσης τις προσωρινές θέσεις εργασίας, ένα φαινόμενο που ε, βλέπουμε τώρα στην Ιρλανδία. Έχουμε υποβάλει λοιπόν τις προτάσεις μας στην Κομισιόν, νομίζω ότι θα τις εξετάσουν. Το βασικό για όλους μας όμως είναι τι ακριβώς θα κάνει η Ευρώπη στην περίπτωση των ε, δικτών που δεν φτάνουν τα επίπεδα αναφοράς. Δεν θα πρέπει να είναι μια ανώδυνη προσπάθεια αυτή, πρέπει να δούμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση ε, ε, που μας αναφέρετε τι κάνετε στη δική σας βολή. Ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον κύριο Γκεντίνη που είναι... Α, κυρία, συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος από την Ιταλική Γερουσία, το Δημοκρατικό Κόμμα, Παρτί του Δημοκρατικού. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα, για να εξοικονομήσουμε και χρόνο. Θέλω να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την δική σας εισήγηση και την ε, παρέμβαση, την ομιλία της κυρίας Ορουά με τις ιδέες που περιελάμβαναν. Η εισαγωγή κοινωνικών δικτών που στη συνέχεια μπορεί να βελτιωθεί, ε, να καλυφθεί καλύτερα, είναι πολύ σημαντική. Δεν πρέπει να προβλέψουμε ουδέτερους δείκτες, αλλά πραγματικά να δούμε θέματα ευαίσθητα όπως η ισορροπία μεταξύ των φύλων ή πώς εκπροσωπούνται οι διάφορες ηλικιακές ομάδες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, να αποτιμήσουμε σωστά τον αντίκτυπο της κρίσης και να δούμε κατά πόσον όντως επιτυγχάνεται η ε, σύγκληση ανάλογα με το φύλλο ή με τις διάφορες ηλικιακέ ομάδες. Πρέπει να εργαστούμε με ταχύτητα για να μπορέσουμε να προβλέψουμε τους κατάλληλους δείκτες και αυτό ε, άμεσα ώστε να ορίσουμε οικονομικές και μακροοικονομικές στρατηγικές προκειμένου οι προσπάθειες για τη μικροοικονομική σταθεροποίηση και την ε, εξυγίανση των προϋπολογισμών να λαμβάνουν υπόψη και τις κοινωνικές ε, πτυχές. Δηλαδή να είναι όλα αυτά βιώσιμα για την ποιότητα ε, ζωής, για το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και για μία ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη. Πραγματικά Ελπίζω η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να καταλαβαίνουν ότι για την εισαγωγή κοινωνικών δικτών θα πρέπει να προβλέψουμε και κοινωνικά μέτρα στις διάφορες οικονομικές συμφωνίες, στα σύμφωνα σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Αναρωτιέμαι μήπως μπορούμε ευθύ αμέσω να δούμε τις κοινωνικές πολιτικές δράσεις, όπως το πρόγραμμα εγγύηση για τους νέους. Μήπως αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε με τρόπο διαφορετικό, ανάλογα με τις οικονομικές ισορροπίες που διαμορφώνονται και τους οικονομικούς δεσμούς που οι διμερείς συμφωνίες, οι συμφωνίες σε επίπεδο ένωσης μπορεί να επιβάλλουν. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στο ο Ρίχαρτ Φάιλου για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα ε, να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της ελληνικής προεδρίας, αλλά θα ήθελα λίγο να σας προειδοποιήσω, μην τρέφετε πάρα πολλές αυταπάτες για το Αρινό Συμβούλιο, αν δεν καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε αυτή την κοινωνική διάσταση, σε όλα τα κράτη-μέλη θα υψωθούν φωνές ότι α, είναι θέμα επικουρικότητας, είναι θέμα παραδόσεων. Ε, εάν το εντάξουμε. Αν δεν το εντάξουμε στο Ερεινό Συμβούλιο δεν θα προχωρήσουμε πουθενά. Θυμάστε τη στρατηγική της Λισαβόνας ε, και το σύνθημα καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας και πού καταλήξαμε λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη απασχόληση συνεχώς. Και αν το αφήσουμε στα χέρια των κρατών μελών δεν θα είναι καθόλου θετικό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομος και σαφής υπήρξατε. Ε, θα δώσουμε τώρα το λόγο ε, σε κάποιον από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ε, της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι η κυρία Σκέβη Κουκούμα. Α, κυρία Πρόεδρε. Η κυπριακή εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος μνημονιακής συναντήληψης είναι πικρή Δεδομένου ότι η μονολυθική πολιτική λιτότητα που έχει επιβάλει η Τρόικα μέσα από του σκληρού όρου και πρόνοια του μνημονίου στερείται προοπτικών ανάπτυξη που λογικά θα, θα έπρεπε να αποτελούσε προπόθεση για έξοδο από οποιαδήποτε οικονομική κρίση. Οι πρωτοφανεί αποφάσει του Eurogroup τη 15η και 25η Μαρτίου για την απομείωση των κυπριακών καταθέσεων έχουν οδηγήσει την κυπριακή οικονομία σε φαύλο κύκλο ύφεση έχουν συμβάλει στην παράλυση του χρηματοπιστωτικού του συστήματο σε μια νύχτα, έχουν διευρύνει τα επίπεδα τη μαζική φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν οξύνει τα επίπεδα τη ανεργία, καταγράφοντα τη ψηλότερη αύξηση ποσοστού ανεργία στην Ευρωζώνη και έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Να πω μόνο ότι η ανεργία από το 4% βρέθηκε στο 17,3% με το 38,5% να είναι νέων. Η μείωση των μισθών μέχρι τέλος του 2014 υπολογίζεται να είναι κατά 30% λιγότερο, με αγοραστική δύναμη να ανέρχεται στην εποχή του 1995. Κατοικίες οδηγούνται σε εκποιήσεις και σύντομα θα βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο των αστέγων. Ε, συμφωνώ με την πρόταση να προσθεθούν και άλλοι δείχτες και είναι γεγονός ότι θα πρέπει να μελετήσουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δείχτες. Ε, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στήριξη των ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού, να επικεντρωθούμε ω πολιτεία στην καταπολέμηση τη ανεργία αλλά και ω Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην παραγωγική δραστηριότητα, την προστασία τη εργασία και των σεβασμών των εργασιακών θέσμιων και του μοντέλου εργασιακών σχέσεων, το οποίο βασίζεται στην κοινωνική διαβούλευση και των θεσμών των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων, όπω έχετε αναφέρει και εσεί, κυρία Πρόεδρε, και την ανασυγκρότηση τη κοινωνική πολιτική με στόχο τη δικαιότερη ανακατανομή του εθνικού εισοδήματο, την καταπολέμηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Και τώρα το λόγο έχει για δύο λεπτά ο συντονιστής ε, των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Απασχόλησης, ο κύριος Αλεχάνδρο Θέρκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ καλωσορίζω τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Προσωπικά φρονώ ότι εκεί πραγματικά θα δοθεί η μάχη για το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ας μην γελιόμαστε. Η κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό μοντέλο ήταν πάντα ο φτωχός συγγενής των κοινοτικών πολιτικών. Ήταν μια πολιτική απλώς αποτελεσμάτων που είχε υποταγή απλούστατα στην οικονομική ε, πολιτική. Και στην ηρωική εποχή Ντελόρ ψηφίστηκαν πάρα πολλοί νόμοι που σήμερα μετά τη διεύρυνση και την ηγεμονία των φιλελεύθερων ιδεών δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο ε, από τη σκληρή νομοθεσία αν μη τι άλλο. Και ο συντονισμός έχει δείξει ε, ποια είναι τα όρια του, ποια ε, είναι η δυσκολία όταν ε, γίνεται μία μάχη για την παγκοσμιοποίηση, ένα ντάμπινγκ προς τα κάτω, μία κούρσα για τη μείωση των μισθών και των κοινωνικών προδιαγραφών και προτύπων. Είναι καθημερινό φαινόμενο. υπάρχει ανάγκη λοιπόν αύξηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, αναβάθμιση του ρόλου της Ευρώπης παγκοσμίω και μαζί με την οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνήσεις ότι δεν νοείται οικονομική διακυβέρνηση χωρίς κοινωνική διακυβέρνηση. Επίσης καταλάβαμε επιτέλους ότι δεν μπορεί να υφίσταται νέο νόμισμα χωρίς ενιαία οικονομική πολιτική. Δεν αρκεί όμως ούτε εσωτερική αγορά ούτε οικονομική πολιτική χωρίς συγκρίσιμες κοινωνικές προδιαγραφές. Αλλιώς θα σπάσει η Ευρώπη σε Ευρώπη δύο ταχυτήτων, την Ευρώπη της ανεργίας από τη μια και την Ευρώπη ε, της φτηνής εργασίας από την άλλη. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν είναι μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά θα πρέπει να σώσουμε και τις επιχειρήσεις μας και ε, μάλιστα το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο σε κάποιον από τη Φιλανδία, Αρκ Γιάλονεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την τελευταία εβδομάδα ακούσαμε πολλές ομιλίες. Σε πολλές από αυτές ελέγχθη ότι η Ευρώπη έχει ξεπεράσει την κρίση, αλλά έχουν γίνει πολλές περικοπές, υπάρχει μεγάλη ανεργία και φτώχεια. Αν δούμε το παράδειγμα της Ελλάδας, απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. υποβάλλονται αιτήματα βοήθειας, στήριξης, ε, αλλά θα πρέπει να συνδέονται αυτά με κάποιες προϋποθέσεις. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον χωρίς ε, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση σε αυτά τα προβλήματα όσο γίνεται πιο σύντομα, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα κοινωνικά προβλήματα. Και η ανεργία εξαπλώνεται στην Ευρώπη και για να ξεφύγουμε από αυτήν θα πρέπει να φροντίσουμε να λάβουν επαρκή υποστήριξη τα κόμματα που είναι υπέρ της Ευρώπης στις επόμενες ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Απασχόλησης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τόμας Μάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι. Την περασμένη εβδομάδα Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό σας, τον κύριο Σαμαρά, στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Εδώ κάθομαι κύριε Βρούτση. Και ε, νομίζω ότι ήταν ε, πολύ ε, ωραία ομιλία του. Ήταν και πρώην συνάδελφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κύριος Σαμαράς. Μας είπε πολύ ενθαρρυντικά πράγματα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε η κρίση έδειξε την αντίφαση μεταξύ του ε, ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που δεν έχει υλοποιηθεί και ε, ανάμεσα στις μεγαλόστομες δηλώσεις της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Στη χώρα σας έχουν γίνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το έχει επιβεβαιώσει όσα άλλοι το αμφισβητούν. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτές οι επιτυχίες στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να γίνουν γνωστές και σε άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν ε, γίνει έλεγχος τώρα από την Τρόικα, την οποία βλέπει με πολύ επικριτικό μάτι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί χρειάζεται δημοκρατικός έλεγχος. Η δυνατότητα ε, αυτή άμεσης επέμβαση τη Τρόικα δεν είναι σημαντική προϋπόθεση. Δεύτερον, μιλήσατε για την ανεργία των νέων. Έχουμε 6 δισεκατομμύρια ε, ως ε, πρώτο σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και το θεωρώ σημαντικό. Αυτό έχει επιπτώσεις. Γίνονται αισθητέ αυτές στη χώρα σας, στη Γερμανία. Ε, έχουμε έλλειμμα ειδικευμένων εργαζομένων και θέλουμε να προσελκύσουμε εργαζόμενους για, για να βγούμε από την ανεργία, όχι για να υπάρξει διαρροή εγκεφάλων από τις χώρες. Αυτό είναι γνωστό. Και επίσης πώς αντιμετωπίζετε τους ενδεχομένους εξτρεμιστές ακραίους ε, εξ αριστερών και δεξιών που ενδεχομένως μπορεί να έχουν και επιτυχίες στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε σε αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά ε, μετά το τέλος το, ε, της σημείωσης των ε, ομιλητών. Έχουμε άλλους τρεις. Να ακούσουμε άλλους ομιλητές. Ο Γκουστεν Μίζελο από την Πολωνική Γερουσία και ζητώ συγγνώμη που μάλλον κατακρεούργησα το όνομά σας. E, Κυρίες και κύριοι, η Πολωνία εξετάζει με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πολωνία δεν ανήκει στην Ευρωζώνη και δεν χρειάστηκε να μεταρρυθμίσουμε τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, διότι το κάναμε αυτό με συστηματικό τρόπο και έτσι καταφέραμε να αποφύγουμε αυτήν την τόσο έντονη κρίση. Ωστόσο, έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Φοβόμαστε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε νέα κριτήρια για την προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Φοβόμαστε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε Ευρώπη δύο ή και τριών ταχυτήτων. Και υπάρχει και η ανησυχία μήπως ε, κατά πόσο βρισκόμαστε ακόμα εντός των πλαισίων ε, της συνθήκης μας. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να γίνουν αποδεχτές από την Πολωνία υπό την προϋπόθεση να πρόκειται για στοχευμένα μέσα και οι συστάσεις να είναι σαφείς και επικαιροποιημένες. εάν διευρυνθούν και αν ε, οδηγηθούμε σε σύγκληση σε κάποιους τομείς, ε, φοβούμαστε ότι αυτό θα επιδεινώσει την ανταγωνιστικότητά μας και αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Γι' αυτό από τη μία εξετάζουμε την πρωτοβουλία αυτή με πολλές ελπίδες, από την άλλη Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Επί της αρχής η Πολωνία πάντως θέλει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ. Ο Φιλίπ Πουλό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μου φαίνεται προφανές ότι πρέπει να ενταχθεί και μια κοινωνική διάσταση στην ΟΝΕ. Αλλά παρόλο που πρόκειται για κάτι το αυτονόητο, βρίσκω ταυτόχρονα ότι δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Θα μπορούσαμε πραγματικά να στοχεύσουμε και να επεξεργαστούμε καλύτερα την προοπτική αυτή που θα επέτρεπε μια μεγαλύτερη σύγκληση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον αριθμό των ε, δικτών στον πίνακα αποτελεσμάτων, δείκτες που τους θέλουμε υποχρεωτικούς και δεσμευτικούς. Παρομοίως, πιστεύω, ότι θα πρέπει να δράσουμε και σε νομοθετικό επίπεδο και στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Βρισκόμαστε σε μία κοινωνική οικονομία των αγορών. Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές, αλλά να έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της σύγκλησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη δέσμευση, ως προς να έχουν μεγαλύτερη δέσμευση μάλλον οι επιχειρήσεις ως προς την κοινωνική τους ευθύνη. Θα πρέπει και να δράσουμε και να αναλάβουμε λοιπόν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη, στο επίπεδο των επιχειρήσεων και έτσι θα επιτύχουμε καλύτερη κοινωνική σύγκληση. Σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων επίσης, Νομίζω ότι βλέπουμε ξανά ποια είναι τα όρια της επικουρικότητας. Ίσως στο Ευρωκοινοβούλιο να το συνειδητοποιούμε πολύ περισσότερο από ό,τι στα εθνικά κοινοβούλια. Εκεί ίσως χρειάζεται λίγη περισσότερη Ευρώπη, αλλά καταλαβαίνω ότι οι εθνικές αρμοδιότητες, οι εθνικά προνόμια δεν μπορούν να θυγούν, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε μηχανισμούς κοινωνική σύγκληση τέτοια, που να είναι δεσμευτική τουλάχιστον ε, η στόχη και να υπάρχει μια ε, προσπάθεια με ανατομέα να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά, να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό dumping και να ικανοποιήσουμε και τα οικονομικά κριτήρια αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες. Ευχαριστώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Καριμαντελή, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλοι οι παρόντες συμφωνούμε λέγοντας ότι θα πρέπει η κοινωνική πτυχή να προσθεθεί στην ΟΝΕ. Ωραία. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Πέντε χρόνια τα λέμε αυτά. Και μετά από μία πενταετία έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η κοινωνική διάσταση εξακολουθεί να μην είναι προτεραιότητα ούτε στο Συμβούλιο ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε έτσι ώστε αυτή η κοινωνική διάσταση της ε, ΟΝΕ να καταστεί πραγματική προτεραιότητα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ερώτηση δεύτερη σε σχέση με τη δική σας έκθεση κυρία Μπερές μας έκανε μια καταπληκτική έκθεση και παρουσίασε η κυρία Βερές ότι αυτή η κρίση χρειάζεται αντιμετώπιση οικονομική και χρηματοπιστωτική. Και ήδη τότε λέγατε στην έκθεσή σας πριν από λίγα χρόνια, Πρόεδρε, ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πραγματικά μια ευφυή ανάπτυξη ε, στην ενεργειακή μετάβαση, τα είπε θαυμάσια ο υπουργό αυτά, ε, για την καινοτομία, την κοινωνική κτλ. Και εγώ έχω πρόβλημα όμως εδώ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί επίσης να είναι πηγή νέων προτάσεων και στηρίζεται από τα Εθνικά Κοινοβούλια, πώς είναι δυνατόν σήμερα να έρχεται σε αντίφαση ε, με αυτά που αποφασίζει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχω και μια μικρή ερώτηση προς την Ελληνική Προεδρία. Είπατε κάτι κύριε Υπουργέ, ότι εμείς δεν έχουμε μαγικές λύσεις για την ανάπτυξη. Περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη, δεν έχουμε καμιά μαγική συνταγή. Μα και πρόσφατα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απεφάνθη ότι δεν θα έρθει ούτε φέτος η ανάπτυξη. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα πούμε στους ευρωπαϊκούς λαούς ότι περιμένουμε την ανάπτυξη με σταυρωμένα τα χέρια ή θα αναπτύξουμε εναλλακτικέ, όπως πρότεινε η κυρία Ουρουά και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καθυστέρηση έχουμε ήδη, δεν υπάρχει θέμα, αλλά επειδή ο Υπουργό προσωπικά ε, ερωτήθηκε δι, θα του δώσω το λόγο για να απαντήσει. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα το μόνο που δεν έκανε ήταν να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Παλέψαμε ως ελληνική κυβέρνηση να αλλάξουμε πολλά στην Ελλάδα και αλλάξαμε και θα εξηγήσω τι αλλάξαμε. Όμως για το θέμα της ανάπτυξης στην εισήγηση που έκανα είπα ότι νικήσαμε για πρώτη φορά τα δίδυμα ελλείμματα αυτό του εμπορικού ισοζυγίου πληρωμών προβλέπεται και μάλιστα κατά ένα χρόνο νωρίτερα ότι το 2014 η Ελλάδα περνάει από την ύφεση στην ανάπτυξη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, εκτός αυτό που είπα, τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Αυτό είναι το οικονομικό αποτύπωμα, η οικονομική επίπτωση των μεταρρυθμίσεων και των πρωτοβουλειών που πήρε η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια και συνεχώς παλεύουμε και δίνουμε τη μάχη για την περισσότερο βελτίωση των, ε, της οικονομίας στη χώρα μας. Στην Ελλάδα. Για τις άλλες ερωτήσεις οι οποίες υπόθηκαν για τις ε, μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να σας πω, και ευχαριστώ για την ερώτηση, ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έγιναν οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πιστέψτε με ήταν και αναγκαίες. Ήταν και αναγκαίες να γίνουν. Γιατί είχαμε διαρθρωτικά προβλήματα αιτία του κακού για την κρίση στην Ελλάδα, μιλάω τώρα μόνο για την Ελλάδα, δεν ήταν μόνο τα διαρθρωτικά προβλήματα, ήταν και γενικά προβλήματα κατασκευαστικά της δομής της Ευρώπης. Αλλά ας πάμε τώρα στην πλευρά της Ελλάδας. Εκεί πράγματι είχαμε διαρθρωτικά προβλήματα. Στην αγορά εργασία είχαμε τρομακτικούς περιορισμούς και τα αλλάξαμε. Πήραμε, είχαμε το πολιτικό θάρρος να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στον κατώτατο μισθό, ως υπουργό έφερα μία μεταρρύθμιση και δημιουργήσαμε πλέον ένα νέο μηχανισμό του μισθού. Ένα μηχανισμό ο οποίος διαμορφώνει το κατώτατο κατόφλι ασφαλεία για όλους τους εργαζόμενου και από εκεί και πέρα ελεύθερα οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να δίνουν οποιοδήποτε μισθό προς τα πάνω. Και ακούστε τι έγινε. Πριν ένα μήνα ανακοινώθηκε η πρώτη κλαδική σύμβαση μεταξύ εταίρων, εργαζομένων και ε, επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα που έδωσε την πρώτη αύξηση μετά από πέντε χρόνια. Άλλη μια θετική είδηση για την Ελλάδα. Η αδήλωτη εργασία ήταν ένα το χειρότερο φαινόμενο. Εργαζόμενοι που δεν δηλωνόντουσαν και πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με ένα σύστημα πρωτοποριακό που το ονομάζουμε Άρτεμις, χτυπήσαμε στη ρίζα του την αδήλωτη εργασία. Βάλαμε το υψηλότερο ιστορικά πρόστιμο που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της χώρας για την αδήλωτη εργασία. Και σήμερα πλέον για πρώτη φορά βλέπουμε μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης. Και αυτό φαίνεται και στα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών που αυξήθηκαν μετά την επιβολή του προστίμου που έδειξε ότι αυτό το πρόστιμο έπιασε τόπο. Άρα σωστή και αυτή η μεταρρύθμιση. Σήμερα το κόστος αναμονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά 21% στην Ελλάδα που, δίνει, που δείχνει ότι αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Έντονα, πολύ ενώ οι πρόβλεψαν για 15% το πήγαμε στο 21%. Όλο αυτό είναι κάτι που τώρα γεννιέται. Και γι' αυτό το 2013 φάνηκε μια ισορροπία στην αγορά εργασίας όσο αφορά την ανεργία. Φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκε, το επαναλαμβάνω. Το δείχνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat. Το τρίτο τρίμηνο ξεκινήσαμε από το 13 27,4% ανεργία, 27,2% και πέσαμε το τρίτο τρίμηνο στο 27% και προβλέπουμε ότι το 2014 θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση. Και επαναλαμβάνω, αξιοποιήσαμε κάθε πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ταμείο το οποίο είναι στο Υπουργείο Εργασίας που έχω την ευθύνη αξιοποίησε και το τελευταίο ευρώ για προγράμματα ανεργίας. Και τα 6 δις ήταν μια καλή εξέλιξη. Τα αξιοποιούμε και τα καταθέτουμε με το Youth Guarantee. Όμως χρειάζονται περισσότεροι πόροι εδώ να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, όλους σας που λάβατε το λόγο στη συζήτηση αυτή. Ε, δεν θα κάνω τώρα τα συμπεράσματα εγώ, διότι στη συνέχεια στην Ολομέλεια θα βγάλουμε τα συμπεράσματα. Ε, ελπίζω ότι θα είμαι Πιστή στα όσα είπατε αναφέροντας τα λεγόμενά σας. Ε, πάντως για το θέμα αυτό ο καθένας έχει την άποψή του. Καλό είναι να συνεισφέρουμε όλοι. Ε, κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι καλή επιτυχία στη συζήτηση στο ΕΠΣΚΟ για ε, αυτό το θέμα του πίνακα αποτελεσμάτων και τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Σας ευχαριστώ. Merci. Λοιπόν, Ευχαριστώ και για τα χειροκροτήματα. Ε, θα παρακαλούσα τώρα ε, τους ε, ομιλητές ε, να αλλάξουμε το πάνελ τώρα γιατί θα πρέπει να καλωσορίσουμε το δεύτερο τμήμα της συνεδρίας. Donc, euh, à la Και καλώ στο βήμα τον κύριο Σαλωμόν αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της Ρουμανικής Βουλής, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακικής Βουλής, τον κύριο Μπλάχα, και τον κύριο Σέρχιο Γκουτιέρης Πριέτο, που είναι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ε, την ανάπτυξη και την κοινωνική της διάσταση. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνονται οι εργασίες. Ε, ευχαριστώ ε, τους ε, τρεις νέους ε, ομιλητές στο πάνελ που ήρθαν στο Προεδρείο. Θα ασχοληθούμε τώρα με τα θέματα απασχόλησης, την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης και σε σχέση με την εγγύηση για την νεολαία και σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς επίσης και το πώς θα κινητοποιείται το νέο πλέον κοινωνικό ταμείο. Τηλεγραφικά θα ήθελα να θυμίσω ότι για την εγγύηση για την νεολαία στο παρόν στάδιο μόλις 17 είναι τα κράτη-μέλη που έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα οριστικά του σχέδια για την υλοποίηση της εγγύησης που κανονικά όμως από 1η Πρώτου 2014 έχει τεθεί σε ισχύ και νομίζω ότι από πλευρά Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της θητείας θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αναχώρα το πώς ευθυγραμμίζεται η κάθε εθνική πρόταση με το πνεύμα ε, της εγγύησης που υποστήριξε πολύ το Κοινοβούλιο αλλά τελικά είναι η σύσταση του Συμβουλίου. Ακόμα και αν επέμεινε πάρα πολύ το Κοινοβούλιο, η εγγύηση αυτή για την νεολαία να έχει αρκετά μεγάλη πρικοδότηση και μάλιστα άμεση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το ίδιο. Και στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την ε, ε, εργασία των νέων που θέλησε να κινήσει το Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτή η ετήσια εξέταση της ε, ανάπτυξης και της μεγέθυνσης οικονομίας τι λέγει. Τα στοιχεία για την ανεργία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη και μάλιστα βαίνουν επιδεινούμενα αυτά εδώ και καιρό. Όχι μόνο για τη συνολική ανεργία, αλλά και ιδιαίτερα για την ανεργία των νέων, τονίζω. Γι' αυτά είναι στοιχεία που δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να αγνοούμε όταν συζητούμε για την ετήσια εξέταση της ανάπτυξης. Υπό την έννοια αυτή, ε, θα αφιερώσουμε το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης και θα ήθελα και πάλι ε, να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου Δημήτρη Κρεμαστινό που είναι πρόεδρος ε, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Βουλής των Ελλήνων. Για πέντε λεπτά παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπέρας για την πρόσκληση. Ε, Βεβαίω ε, θα επαναλάβω και πάλι αυτό που είπα στην προηγούμενη συνεδρία ότι δυστυχώς ε, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ενεργεία των νέων καθώς πλησιάζει το 60% των νέων και ακολουθείται από την Ισπανία. Και πάλι δηλαδή ο Νότος δυστυχώς πρωτοπορεί σε αυτό το θέμα και παρά τα προγράμματα τα, με πολλή επιμέλεια τα οποία έχουν υποβληθεί και εκτελούνται, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Βρούτσης, τα αποτελέσματα είναι ε, πενιχρά, είναι πάρα πολύ αδύνατα. Η προβλεπόμενη καταπολέμηση ενεργείας με αυτό το ρυθμό, στην καλύτερη περίπτωση, ανάγεται σε ποσοστά του 1% ανά έτος. τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ε, τα προσεχή χρόνια ε, μια ολόκληρη γενιά νέων ε, θα ζήσει με την ανεργία και πώς θα αναπτυχθεί οι χώρες όταν οι νέοι, η νέα γενιά μεγαλώσει με την ανεργία. Ποια θα είναι η υποδομή αυτή της γενιάς. Είναι δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ερώτημα α, περίπου υπαρξιακό για τις ίδιες τις χώρες και φυσικά την οικονομία τους. Α, όμως ε, ε, και πάλι θα επαναλάβω αυτό που είπα στην προηγούμενη σέσιο. Χωρίς ε, ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους που να είναι της τάξεως του 3 έως 5% ετησίως του ΑΕΠ πρακτικά είναι αδύνατο να περιμένει κανένας καταπολέμηση της ενεργείας με τα προγράμματα αυτά τα οποία περίπου είναι όπως η ασπιρίνη, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται όχι σαν φάρμακο για να ρίχνει τον πυρετό ή τον πόνο, αλλά για να θεραπεύσει την ίδια την πάθηση. Η πάθηση δεν θεραπεύεται. Τα προγράμματα λοιπόν είναι η ασπιρίνη η οποία χορηγείται για να βελτιώσουμε την κατάσταση, να βελτιώσουμε τη ζωή, αλλά όχι για να λύσουμε το πρόβλημα. Αντίθετα, επαναλαμβάνω, θα περιμένει κανένας από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα τολμηρά προγράμματα στο θέμα που λέγεται ανάπτυξη και χωρίς ε, αναπτυξιακά προγράμματα που θα εξασφαλίσουν ένα ποσοστό γύρω στο 3 5% για χώρες του Νότου ετήσια αύξηση του ΑΕΠ πρακτικά είναι αδύνατο να περιμένει κανένας θεαματικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της ανεργίας. Α, τώρα όσον αφορά το θέμα το συνταξιδοτικό εάν ένας ρωτήσει ότι εάν ε, υποχρεωθεί κάποιος να τιμωρήσει κατά κάποιο τρόπο κοινωνικά τους ανθρώπους και αποφασίσει να μειώσει μισθούς στις συντάξεις αντιλαμβάνεστε ότι ο πιο ευαίσθητος χώρος είναι οι συντάξεις διότι ο νέος μπορεί να απασχοληθεί, να δουλέψει περισσότερο, να δουλέψει περισσότερες από μία δουλειά, Ο συνταξιούχος και ο γέρος δεν μπορεί δυστυχώς να ανταποκριθεί είναι υποχρεωμένος να ζήσει με αυτό που μια ζωή, αν θέλετε, κατέβαλε. Το να μειώνονται λοιπόν οι συντάξεις όπως συνέβη στις χώρες του Νότου είναι περίπου κοινωνικά εγκληματικό διότι αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται αφού προσέφεραν μια ολόκληρη ζωή ε, τιμωρούνται στα γεράματά τους να ζήσουν άσχημα χρόνια. Αυτό το, αυτό το γεγονός αυτό καθεαυτό αυτό δεν συνιστά πολιτισμό, δεν συνιστά χώρες με ψηλό επίπεδο δίχτυ ε, πολιτισμικό. Ε, και η Ευρώπη βέβαια ανήκει σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή στις χώρες που έχουν υψηλό πολιτισμικό δίχτυ. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουν διαφορετικά το θέμα το συνταξιδοτικό. Και έτσι λοιπόν οι διάφορες μεταρρυθμίσεις που σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητιώνται, πρέπει να είναι ουσιαστικές και να κατατείνουν στο να διασφαλίσουν τουλάχιστον το μήνυμο της σύνταξης που θα εξασφαλίσει μια ανθρώπινη ζωή στο συνταξιούχο ο οποίος αν θέλετε είναι αυτός που τελικά τη δικαιούται αφού μια ζωή έχει προσφέρει και έχει δουλέψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε και είναι πολύ σταράτα τα λόγια σας αυτά. Ευχαριστώ ε, για την εισαγωγή της συζήτησης. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντριάν Σόλομον, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ε, της Ρουμανικής Βουλής θα μας μιλήσετε και για τις ανισότητες που αυξάνονται στη Ρουμανία, αλλά και γενικότερα για τα κοινωνικά στοιχεία της ετήσιας εξέτασης ε, της ανάπτυξης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αγαπητέ συνάδελφοι, έχετε το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι βουλευτές, είναι σημαντικό για μένα να μπορώ να συμβάλλω σε αυτήν τη σημαντική συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχω μοιράσει σε τέσσερα μέρη την παρουσίασή μου. Καταρχάς, θα εξετάσω το θέμα της απασχόλησης και θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση του αντικτύπου της κρίσης. Δεύτερον, ε, θα εξετάσω τον ε, έντονο κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης και γιατί διήρκησε τόσο πολύ. Κατόπιν ε, θα εξετάσω την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων που έχουν ληφθεί για να μετριαστούν οι συνέπειες της κρίσης. Και τέλος, θα σας δώσω τη δική μας άποψη σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι τα μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, λοιπόν, κοινωνικός αντίκτυπος ε, της κρίσης. Ε, μπορεί να ε, το χωρίσει κανείς αυτό ως εξή. Υπάρχει υψηλή ανεργία στους νέους, υπάρχουν όλο και περισσότεροι που κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από τα επίπεδα της φτώχειας. Επίσης υπάρχει αυξημένη ανισότητα εντός των χωρών λόγω του ανοίγματο της ψαλίδας των εισοδημάτων. Έχουμε αποδυναμωμένη δυνατότητα ανακατανομής ε, στα συστήματα φορολογίας και κοινωνικής προστασίας. Η ανεργία αυξάνεται, κάτι που επιβαρύνει την αγορά εργασίας και μπορεί να έχει σημαντικό διαφορετικό αντίκτυπο. Κάτι που επίσης ε, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις δυνατότητες ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Είναι λοιπόν ζωφερή η εικόνα της ε, κρίσης και οι προβλέψεις για την απασχόληση είναι επίσης ζωφερές όπως περιγράφονται οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση ανάπτυξης. Λαμβάνεται υπόψη η απόσταση από την ε, κοινωνική αποκατάσταση και ε, δεν αναμένεται να βελτιωθεί η κατάσταση σύντομα και υπάρχουν ε, πολλοί παράγοντες ε, που θέτουν σε κίνδυνο την ιδέα της ελληνικής. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος μεγάλης πολιτικής κρίσης που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική κρίση και η αύξηση των ανισοτήτων ε, είναι κάτι πολύ δυσάρεστο και το οποίο μάλιστα ευνοεί τον λαϊκισμό διότι ζητάτε έτσι η, η πάυση ε, ενός από τα δασκότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της ελεύθερης κινητικότητας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους που αμφισβητούν το δικαίωμα αυτό, διότι είναι ξεροφοβικοί στην ομιλία τους. Δεύτερον, η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την κρίση Ε, είχε να κάνει με ε, την αυτοσυγκράτηση, την, ε, τον τη δημοσιονομική πειθαρχία, την συγκράτηση της, του πληθωρισμού, αλλά η κρίση μας δείχνει ότι η σταθερότητα των τιμών δεν αρκεί για να διασφαλιστεί η μακροοικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, το ίδιο οικονομικό δόγμα που στηρίζεται και από την λεγόμενη ορθοδοξία του Μάστριχτ μας δείχνει ότι η κρίση αυτή θεωρήθηκε κρίση δημοσίου χρέους και όχι ιδιωτικών φορέων. Οι προσαρμογές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με τις οδηγίες του ε, ε, εγχειριδίου οδήγησαν σε στασιμότητα. Και Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ευελιξίας για τις πλεονασματικές χώρες, ε, όχι όμως για τις χώρες που έχουν έλλειμμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα στις χώρες που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους και υπάρχουν φόβοι για αποπληθωρισμό και ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης ε, έχει οδηγήσει σε μία όχι βελτιστή αντιμετώπιση. Είχαμε ε, μεγάλη ύφεση την οποία χειριστήκαμε με χειρότερο τρόπο από ότι την μεγάλη οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930. Περνώ στο τρίτο μέρο τη παρουσίασή μου που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για να μετριαστεί ο αντίκτυπο τη κρίση. Οι πολιτικέ και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για να βελτιωθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη βασίζονται στην ιδέα ότι η ανεργία οφείλεται στην ακαμψία της αγοράς. Έτσι λοιπόν ε, ασχοληθήκαμε κυρίως με την αγορά εργασίας και όχι με τις πολιτικές απασχόλησης. Οι πολιτικές επικεντρώνονται σε διαφορετική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μείωση της κοινωνικής προστασίας, ε, μείωση της, ε, βελτίωση μάλλον του ταιριάσματος ε, δεξιοτήτων και ζήτησης στην αγορά, Επίση, περισσότερη ευελιξία στι συλλογικέ συμβάσει, ώστε να υπάρχει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των ε, μισθών. Και επίσης έγιναν προσπάθειε να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμο στην εργασία. Η Τρόικα, λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ε, και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά το 2011 στη Ρουμανία. Ε, αλλά φαίνεται ότι πνεόμαστε περισσότερο από την ιδέα ότι η μεγάλη κρίση που περνάμε τώρα είναι μάλλον διακοπές για τους εργαζομένους και ότι ε, εάν και πολλά από τα μέτρα είναι αντιεπικοδομητικά βραχυπρόθεσμα, υπάρχουν ε, οι κυκλικοί παράγοντες, έλλειψη της οικονομικής ανάπτυξης. Δεν έχει λοιπόν αυτό να κάνει με διαφορετικά ε, θέματα. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης με καλή βιομηχανική πολιτική. Ε, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά με περικοπή στους μισθούς. Αυτό απλά θα μειώσει τη ζήτηση. Το αυξημένο δυναμικό από πλευράς της προσφοράς θα το νιώσουμε μόνο ε, εάν έχουμε και αυξημένη ζήτηση. Η μεταρρύθμιση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας μπορεί να βοηθήσει τους ε, εργαζομένους να αναζητήσουν εργασία, δεν θα τους βοηθήσει απαραίτητα όμως να βρουν εργασία. μπορεί να αυξηθούν οι αποπληθωριστικές πιέσεις και αυτό είναι επικίνδυνο. Τέταρτον, χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό μοντέλο και οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι και να αναπτυχθεί η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ με την υιοθέτηση του πίνακα αποτελεσμάτων ε, με το επίκεντρο στην κοινωνική κατάσταση και τα μέτρα για να υποστηριχθούν οι πιστώσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι καλά νέα και πιθανότατα να βοηθήσουν την κοινωνική διάσταση. Δεν ε, μας υπόσχονται όμως σταθερή οικονομική ανάπτυξη τι δεν θα τη δούμε εάν δεν ασχοληθούμε με το θέμα της ανεργίας, διότι όλα αυτά αποτελούν ε, απλά ε, κάποιες αναλαμπές ελπίδας σε ένα πολύ ζωφερό περιβάλλον ε, λιτότητας. Πρόσφατα παρατηρήθηκε ότι η πραγματική αιτία της κρίσης ήταν οι ανισότητες στο εισόδημα, κάτι που έχει επιδεινωθεί από την έναρξη της κρίσης. Η ανισότητες ε, οφείλονται στην ε, αποδυναμωμένη ζήτηση, κάτι που έχει οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη και στην φτώχεια. Γι' αυτό η πραγματική πρόκληση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ασχοληθούμε με τις ανισότητες μεταξύ των χωρών και φυσικά ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ανισότητες εντός των χωρών, αλλιώς θα διηγηθούμε σε οικονομική στασιμότητα. Τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα ήταν προς όφελος μεγάλων δανειστών τραπεζών και ανθρώπων που κατέχουν κεφάλαιο στις ε, χώρες ε, και ήταν εις βάρος των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν δεν είναι βιώσιμο. Χρειαζόμαστε διαφορετικό οικονομικό μοντέλο μέσω του οποίου να επιτευχθεί πραγματική ανάπτυξη με, διάφορους, με διάφορες πηγές εισοδήματος, ε, πιο μεγάλους μισθούς και λιγότερες ανισότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσουμε την ε, προτεραιότητα της δημοκρατίας πάνω από την οικονομία και εξυγχρονισμός του κράτους ε, σημαίνει και να ε, το απελευθερώσουμε από την αγορά και να λειτουργεί υπέρ του κοινού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο πειθαρχημένες αγορές, να αποτελούν μέρος της κοινωνίας και να ενεργούν υπό τον δημοκρατικό έλεγχο της κοινωνίας. Συμπεράσματα. Η ένταση και η διάρκεια της κρίσης έχουν ε, επηρεάσει την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, μένει στην ορθοδοξία του Μάστρεχτ και πολλά προβλήματα οφείλονται σε διαφορετικά και όχι ε, συγκυριακά προβλήματα και ο προηγούμενος ομιλητής ε, αναφέρθηκε στο να χρησιμοποιήσουμε παρασεταμόλη για να θεραπεύσουμε τον καρκίνο. Αυτό σίγουρα δεν λειτουργεί. Και για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό πρότυπο, καλύτερες θέσεις εργασίας και μείωση των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λούμπος Βλάχα, πρόεδρο της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Εθνικής Βουλής της, της Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακίας, Ναρόντνα Ράντα. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις εμπειρίες της χώρας σας και τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με το πρόγραμμα εγγύησης για τους νέους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα αυτό και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μερικά στοιχεία για την απασχόληση στην ε, Σλοβακία και τα κοινωνικά μας προγράμματα. Σε μια δεύτερη φάση θα μιλήσω για εναλλακτικέ λύσεις που πιστεύω θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές δυσκολίες ε, και λαμβάνοντα αφορμή, όπω είπε ο Ρουμάνο συνάδελφο, να πω ότι η ενεργεία είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα στη Σλοβακία. 13,5 είναι το ποσοστό αυτή τη στιγμή, ενώ η ενεργεία των νέων αγγίζει το 34%. Εάν μάλιστα υπολογίσουμε και τους φοιτητές, ε, φτάνουμε το 14% ε, για το συνολικό ποσοστό ανεργία στη χώρα. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι προτεραιότητα για μας. Έχουμε ένα εθνικό σχέδιο για την υλοποίηση της εγγύησης των νέων στη Σλοβακία και ήδη έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επιτύχει όμως κάποια πρόοδο στην καταπολέμηση της ενεργείας στη χώρα μας χάρη στα ευρωπαϊκά ταμεία με 17 ε, δις ε, ευρώ για να δημιουργηθούν 7.000 θέσει εργασία ε, σε ένα χρόνο τουλάχιστον. Επιδοτούμε εργοδότες που προσλαμβάνουν ε, νέους εργαζομένους ως τα 29 έτη, οι οποίοι έχουν υπάρξει για ε, μακρό διάστημα άνεργοι. Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην υποχρεώνει τους εργοδότες να υποβάλουν κοινωνικές εισφορές. Επίσης, η εργασιακή μας πολιτική λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται και με ετήσιους δείκτες στην ετήσια, στις ετήσιες αναχώρα εκθέσεις. Ε, επί πολλά χρόνια όμως βλέπουμε η ενεργία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ποσοστά. Ποιοι είναι οι λόγοι. Υπάρχουν κάποια δομικά προβλήματα, διαρθρωτικοί λόγοι στη Σλοβακία που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα, που οι συνέπειε τη κρίση ήρθαν να του επιβαρύνουν. Υπάρχουν τρει βασικοί λόγοι για την ανεργία στη Σλοβακία. Η ανισότητα μεταξύ ε, του εκπαιδευτικού συστήματο και τη αγορά εργασία και για αυτό το σκοπό, για να αντιμετωπιστεί το κενό αυτό, ε, το πρόβλημα αυτό, προβλέψαμε διάφορα μέτρα σωστή ενημέρωση των φοιτητών σε επίπεδο πανεπιστημίου για το ποιε είναι οι ανάγκε τη αγορά εργασία, οι πραγματικέ ανάγκε. Επίση, θελήσαμε να έχουμε την απόκριση των φοιτητών, γνωρίζοντα τι πρακτικέ του εμπειρίε και να προσαρμόσουμε ανάλογα την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Άλλοι λόγοι για τα υψηλά ποσοστά ανεργία στη Σλοβακία είναι ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού συγκεντρώνεται γύρω από την πρωτεύουσα της Μπρατισλάβα. Εκεί όμως η ενεργεία των νέων φτάνει το 17,5%. Στο ανατολικό τμήμα της Σλοβακίας φτάνει το 43%. Αυτό είναι καταστροφικό. Γι' αυτό η Σλοβακία χρειάζεται πραγματικά τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία και τα κονδύλια τη ε, της κοινωνικής Διότι οι περιφερειακές ανισότητες στη Σλοβακία είναι ένα πρόβλημα ευρύτερο. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη υποδομών, λόγω χάρη. Η Σλοβακία χρειάζεται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά χρειάζεται και καλύτερη ενσωμάτωση του πληθυσμού των Ρωμά που αποτελούν το 7,5% του πληθυσμού της χώρας, στα ανατολικά κυρίως, και βεβαίως ε, με υψηλά ποσοστά ενεργείας και εκείνη. Ο τρίτος λόγος είναι πολιτικός η ε, πολιτική αστάθεια και η υψηλή ανεργία έχουν να κάνουν με τις ε, κακές ε, κοινωνικές πολιτικές του παρελθόντος με χαμηλό εργασιακό κόστος ως πρώτο στόχο την, ε, τις και τις απολύσεις εργαζομένων. Από το 2004 η Σλοβακία έπρεξε ένα καλό παράδειγμα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου με χαμηλή φορολόγηση των εταιριών, με ε, για υποβολή ποσών, με ιδιωτικοποίηση του συνταξιδοτικού μας συστήματος, στοιχεία που έχουν ήδη μεταρρυθμιστεί από καιρό και βεβαίως με πολλά πλεονεκτήματα προς τους εργοδότες και όχι τους εργαζομένους. Αυτά για να δημιουργήσουν εργοδότες νέες θέσεις εργασίας. Κι όμως αυτό δεν έγινε, γι' αυτό και τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν υψηλότατα στη χώρα μας. Η διαλεκτικότητα και η ευελιξία είναι η πρώτη αντίδραση που θα έπρεπε να έχουμε, ιδίω για να αντιμετωπιστούν οι κερδοσκόποι και όσοι εκμεταλλεύονται το φθηνό εργατικό δυναμικό. Ε, Σλοβακία θα μπορούσε να γίνει ε, αντίληπτη ως, ε, θα μπορούσε να ειδωθεί και ως ένα παράδειγμα αποτυχίας του νεοφιλελεύθερου μοντέλου λόγω και της κοινωνικής κατάστασης και όχι των οικονομικών στοιχείων τα δεν γίνονται μόνο για λόγους ιδεολογικούς. Θέλουμε να διασωθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στηρίζοντας ακόμη τους νέους. Πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κοινωνικής οικονομίας, κάτι που ούτως ή άλλως αναφέρει και νέα πράξη για την αγορά και στην πρώτη και στη δεύτερη εκδοχή της. Πρέπει να προωθηθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Σλοβακία τώρα μόλις αρχίζει να αξιοποιείται προκειμένου να ε, προωθηθεί το επιχειρήν προς όφελος των ε, περιοθυροποιημένων ομάδων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Ρωμά. Έπειτα χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους συνεταιριστικούς οργανισμούς. Αυτό είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη, διότι μπορεί να υπάρξει μια δικαιότερη κατανομή ε, του εισοδήματος και μπορούν οι εργαζόμενοι να συναποφασίζουν και να συντονίζουν οι ίδιοι την παραγωγικότητα. Ε, είναι όλα αυτά στα χέρια των εργαζομένων. Θέλω λοιπόν να απευθύνω έκκληση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να στηρίξουν περισσότερο τις συνεταιριστικού οργανισμούς θέσεις εργασίας που δημιουργούνται έτσι είναι πιο σταθερές. Επίσης πρέπει να δώσουμε έμφαση στα πανευρωπαϊκά κοινωνικά ωφέλη, ωφελήματα κυρίως για τους φτωχότερους. οι κοινωνικές ε, λειτουργίες που πρέπει να καλυφθούν ε, είναι πολλές και Εάν δεν τις λάβουμε υπόψη, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο. Η ιδιότητα του πολίτη, όπως αναφέρεται στη συνθήκη του Μάστριχτ, προβλέπει όχι μόνο πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά και κοινωνικά. Κοινωνικά όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό. Γι' αυτό είμαι πεπισμένο ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και τις συνθήκες εφόσον χρειαστεί, προκειμένου η ευρωπαϊκή ηθαγένεια να είναι κάτι που θα καλύπτει περισσότερες πτυχές. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει για κάποιο είδους επίδομα ανεργίας. Γι' αυτό Μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιδέα του κατώτατου μισθού. Παρόμοιες προτάσεις έχουν υποβληθεί από τον κύριο Σμιτ, ο οποίος μιλά και για ευρωπαϊκές υποτροφίες, αλλά και για τα κοινωνικά ωφέλη που θα πρέπει να καλύπτουν όλοι οι εργοδότες. Το δεύτερο λοιπόν πρόγραμμα που προτείνω είναι η καταβολή κοινωνικών ωφελημάτων προς τους εργαζομένους και δημιουργία μιας κοινωνικής ένωσης. Να υπάρχουν επιδόματα εφόσον χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι αυτό που ε, εδώ καταγγέλουμε δεν είναι η παγκοσμιοποίηση, αλλά το κοινωνικό μοντέλο που δημιουργείται μέσω της παγκοσμιοποίησης. Αυτό το προωθούν οι πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες προάγουν μόνο τα οικονομικά τους συμφέροντα. Υπάρχει πίεση για χαμηλότερη φορολογία με, την, ε, με σε ένα πιο αδύναμο πολιτικό σκηνικό. Αυτό συμφέρει τις εταιρείες, αλλά εμείς δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τα κοινωνικά πρότυπα και την κοινωνική προστασία των πολιτών μας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ε, ανταγωνιστεί τη Λατινική Αμερική, την Κίνα με τις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών. Θέλουμε οι εργαζόμενοι μας να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα με 15 λεπτά του ευρώ αμοιβή την ώρα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας για τον 21ο αιώνα. Θέλουμε να βελτιώσουμε και να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο Δεν θέλουμε περαιτέρω στρέβλωση των προτύπων στον τομέα αυτό και για να ανακεφαλαιώσω η Σλοβακία καταπολεμά την ανεργία όμως το νεοφιλελεύθερο μοντέλο δεν φαίνεται να έχει επιτύχει ε, στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις να πιεστούν, να ασκηθεί πίεση στις κυβερνήσεις για να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανισότητες. Η κοινωνική πτυχή πρέπει να ενσωματωθεί στις οικονομικές πολιτικές. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε την ε, τα κενά των, και τις ε, αποτυχίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και έτσι θα γίνει η Ευρώπη πιο δημοκρατική. Ναι, Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Λέξη δεν είπατε για την εγγύηση για την νεολαία, αλλά ήταν ε, μια θερμή τοποθέτηση δική σας άποψη ε, για τα κοινωνικά ζητήματα. Βεβαίως μπορεί πλήρως να αξιοποιηθεί, είναι η δική σας μάτια. Θα δώσω το λόγο τώρα ε, στο τελευταίο μιλητή. Θα είμαι πολύ πιο αυστηρή για το χρόνο. Δέκα λεπτά και θα σκόψω το μικρόφωνο. 14 ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Κλείνει εδώ ο κατάλογος προφανώς. Ε, Σέρχιο λοιπόν Γκουτιέρης το έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε μένα επισοκλήρως να παρουσιάσω την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα ψηφίσουμε ακριβώς αύριο. Είναι μια έκθεση η οποία έχει το νόημα να προσπαθήσει να φέρει στο ίδιο επίπεδο με τα οικονομικά και τα νομισματικά και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τα θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων για το συντονισμό τους. Έχουμε ένα πλαίσιο γνωστό, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη και κάποιοι ηγέτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν βουλευτές που θέλουν πολύ γρήγορα να έρθει η ανάκαμψη ε, και η ανάπτυξη εξαγγελιών. Μπορεί να υπάρχουν ε, έτσι, ενδείξεις στη μακροοικονομία, στα πρωτογενή πλεονάσματα, στα ισοζύγια τρέχουσών συναλλαγών, στις εξαγωγές, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία ε, και κάποιοι άλλοι που είναι πιο επικριτικοί και μεταξύ αυτών είμαι και εγώ για μικρή βελτίωση μπορεί να υπάρχει στη μακροοικονομική πτυχή, αλλά έχουν γίνει δραματικές θυσίες και έχουν πέσει στο βωμό όλο αυτό οι περισσότερες κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής 2020. Μιλούμε για ανάκαμψη, για ανάπτυξη με 0,0% και 27 εκατομμύρια είναι σχεδόν οι άνεργοι. Ένα στου πέντε νέου στην Ευρώπη παραμένει άνεργος. Σε κάποιες χώρες ε, είναι μέχρι και 50 και 60% η ανεργία των νέων. Σε όλες τις χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται ο κοινωνικός αποκλεισμό καθημερινά και σε όλες τις χώρες επίσης τα νοικοκυριά ε, φτωχαίνουν. Και ιδιαίτερα το θέμα της παιδικής φτώχειας αυξάνεται μήνα με το μήνα. Και αν δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον, θα πρέπει να λέμε και τα δύο. Ναι, εντάξει, συμφωνώ, ε, μακροοικονομικά στοιχεία βελτιώνονται, αλλά υπάρχει και ένα τίμημα εδώ. Ε, ε, θυσιάζουμε πολλέ από τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση αν δεν θέλουμε να κοροϊδευόμαστε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ορισμένοι προσπαθούν να μα πείσουν ότι κερδίζουμε μια μάχη βραχυπρόθεσμη με τα μακροοικονομικά, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κοινωνικά στοιχεία θα επιδεινωθούν και θα είναι σοβαρό πρόβλημα για την αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη και μεσοπρόθεσμα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και το χειρότερο, νομίζω το είπε ο κύριος Σαλωμών, μπορεί να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη, αλλά είναι πιο βραδία από εκείνη που είχε προβλεφθεί στην αρχή και βαθύτατα ανισότητα τα επικρατεί και διάσταση, όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών. Πέρυσι πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά από την ίδρυση των Ταμείων Συνοχής η συνοχή μεταξύ κρατών μελών δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε. Και επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι αυτό μόνο μεταξύ διαφόρων κρατών αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μεταξύ των διαφόρων πολιτών αυξάνονται οι ε, ανισότητες με τρόπο θεαματικό τα τελευταία χρόνια. Εμείς τη ζητούμε στα πλαίσια αυτών των δεδομένων στην έκθεση της οποίας είμαι εισηγητής. Κάνουμε πρώτα μια κριτική ανάλυση. Πώς φτάσαμε ως εδώ. Ας πούμε, να ότι εσφάλαμε, ότι κάναμε λάθος στην οικονομική στρατηγική που υιοθετήσαμε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ε, είχαμε ε, υπερβολική εξυγίαση των προϋπολογισμών ε, δεν λάβαμε υπόψη τους πολλαπλασιαστές ε, στη δημόσια δαπάνη, δηλαδή όσο μεγαλύτερες περικοπές τόσο βαθύτερη ύφεση και τόσο ε, μεγαλύτερες οι κοινωνικές επιπτώσεις. Επιπλέον απέτυχε και το εξής γεγονός. Δεν καταφέραμε να προβλέψουμε τους περιορισμούς που θα γι' αυτό, όχι μόνο για την κοινωνία και για την οικονομία. Οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις μείωσαν την εσωτερική ζήτηση με τη συμπίεση των μισθών με την ανεργία. Δραστικά μειώθηκε σε πολλά κράτη-μέλη ε, το επίπεδο αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Οπότε, ε, όπως λέγω, κάνουμε στην έκθεσή μας αυτή την κριτική ανάλυση. Στη συνέχεια, τι προτείνουμε τώρα. Πρώτον, μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση σε όλη τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μπορεί τώρα να έχουμε φτάσει σε μια διαδικασία που εκχωρείται ε, πολύ κυριαρχία από τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν σε όλες τις αποφάσεις θα πρέπει να εγγυηθούμε να υπάρχει πάντα από πίσω δημοκρατική νομιμοποίηση. Τι σημαίνει αυτό. Όταν γίνονται τα εθνικά σχέδια για τη σταθεροποίηση και τη σύγκληση, τα κράτη-μέλη πριν τα στείλουν στις Βρυξέλλες θα πρέπει να περάσουν από κοινωνικό διάλογο και από εθνικό κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εγκρίνονται τέτοια σχέδια και μετά και το six pack, τα ξέρετε αυτά με τις ε, έξι οδηγίες που είναι και δεσμευτικές, δεν μπορούν όλα αυτά να γίνονται ερήμην των ε, εθνικών κοινοβουλίων που είναι η έκφραση της εθνικής κυριαρχίας. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει συναπόφαση. Εδώ εμείς είμαστε το θεσμικό όργανο που έχει τη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν είμαστε απλό συμβουλευτική συνέλευση. Ε, επίσης όλοι θα πρέπει να συναποφασίζουμε για αυτά τα θέματα. Κάτι άλλο ακόμα που ζητούμε στην έκθεση. Συμφωνούμε βέβαια ότι δεν θα πρέπει να πέσουμε σε αυτή την κόποση των μεταρρυθμίσεων για την οποία τόσο πολύ ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως να είμαστε απαιτητικοί όταν ζητούμε τα διάφορα ε, εργαλεία να εφαρμόζονται για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, αλλά αναζητώντας την ανταγωνιστικότητα δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε στη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω με δραματικές περικοπές. Ε, ούτε μπορούμε να βασιστούμε στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, να πεταχτούν δηλαδή εκατομμύρια εργαζομένων εκτός συμβάσεων, ούτε να κάνουμε εκπτώσεις στις κοινωνικές μας εγγυήσεις. Γιατί οι πολίτες το αισθάνονται αυτός βαθιά αδικία. Δεν φτάνει που χάνεις τη δουλειά σου, δεν φτάνει ε, που ε, είσαι άνεργος. Υπάρχουν ε, εναλλακτικέ λύσεις, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να μας δώσουν παραδείγματα για την ανταγωνιστικότητα. Κοιτάξτε τη βαθμολόγηση, το ranking, ποιες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες είναι ανταγωνιστικές και τι επικρατεί εκεί από εργασιακά δικαιώματα και κοινωνικές συνθήκες. Λοιπόν, αν θέλουμε να προωθήσουμε μια στρατηγική θα πρέπει να έχουμε παραγωγικές επενδύσεις, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερε δυνατότητες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ζητούμε λοιπόν στην έκθεσή μου ένα σύμφωνο για την βιώσιμη ανάπτυξη, για τις συλλογικέ συμβάσεις και για τον ανταγωνισμό, χωρίς αυτό να σημάνει ε, εκπτώσεις, επαναλαμβάνω, στα εργασιακά δικαιώματα και στις συνθήκες. Ε, θέλουμε και μια στρατηγική πιο φιλόδοξη για την εργασία των νέων και όχι μόνο των νέων και των μεγαλύτερων άνω των 45 ετών γιατί πολλές φορές τους ξεχνούμε αυτούς στην κρίση. Και στην εγγύηση ε, για την απασχόληση εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Απασχόλησης ήμασταν πάρα πολύ φιλόδοξοι. Ζητήσαμε μια ευρωπαϊκή εγγύηση, όχι απλώς χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων αλλά μια ε, μεγάλη πολιτική. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της κρίσης 500 δις ευρώ δώσαμε για να σώσουμε τα χρηματοπιστωτικά συστήματα στην Ευρώπη. Τι καταφέραμε για την επόμενη επταετία για ε, την εγγύηση για την νεολαία. 9 δισεκατομμύρια για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία. Ε, μα αυτό δεν είναι ανισορροπία, δεν είναι σημαντική ε, στρεβλή ε, αντίληψη για το ποιες είναι οι προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλους μας απασχολεί και μας ανησυχεί η ανεργία των νέων. Ακούμε για χαμένη γενιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αντιστοιχεί αυτό με τη χρηματοδότηση που προβλέπουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Σαλωμών, καμιά φορά έχουμε την αίσθηση ότι δίνουμε ασπιρίνη για κάταγμα ας πούμε. Όχι μόνο αυτό, καμιά φορά έχεις κάταγμα, δίνεις ασπιρίνη και του λες πάσε και το χέρι σου τώρα γιατί δεν μου φτάνει το πόδι. Ε, αυτή λοιπόν η εγγύηση για την νεολαία και η εξυγίαση του προπολογισμού τι σημαίνει. Στην Ισπανία τις αναλογούν περίπου για 7 ε, χρόνια ένα δισεκατομμύριο. Αλλά ακριβώς λόγω των περικοπών και της εξυγίασης ε, κόβουμε δισεκατομμύρια από την ανάπτυξη. Δηλαδή δίνουμε με το ένα χέρι 300 εκατομμύρια το χρόνο και από την άλλη ε, κόβουμε 5 δισεκατομμύρια για την ανέργεια των νέων από τις εθνικές πολιτικές. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και πολύ πιο προσεκτικοί με τις προτεραιότητες που βάζουμε σε πολιτικό επίπεδο. Και ένα τελευταίο. Θα πρέπει να ανοίξει συζήτηση και για άλλα ευρωπαϊκά μέσα και εργαλεία. Να ανοίξει συζήτηση, διαβούλευση χωρίς φόβο και πάθος, ούτε είναι δεδομένο το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα. Για τους ε, αυτόματους σταθεροποιητές, η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, πέρασε το δεκάλεπτο. Ορίστε, τι να κάνω τώρα, έχω και την πρόοδο. Ε, ε, ε δεύτερα. Ε, ε, έλεγα για τους αυτόματους ευρωπαϊκούς σταθεροποιητές. αν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης είχαμε ένα επίδομα ανεργίας με μια διασύνδεση ένα 1,2% των συνεισφορών ετησίως να μπαίνει σε ένα ευρωπαϊκό κορβανά, ε, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτή τη δραματική αύξηση της ανεργίας. Θα ήταν ένα εργαλείο αλληλεγγύης σε ε, τέτοιες καταστάσεις και σίγουρα ε, θα είχε αποφύγει κάπως την αύξηση των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Συγγνώμη, σας είπα ότι έχουμε 14 ομιλητές. Έχουμε 7 όμως και θα χρειαστούμε 14 λεπτά. Έχει κλείσει ο κατάλογος των αγορητών. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας πρώτα απ' όλα τους τρεις συμμετέχοντες στο πάνελ με την ε, παρουσία του Έλληνα συναδέλφου. Τους ευχαριστώ λοιπόν για τις ομιλίες τους, παρόλο που δεν έγινε πολύ λόγος ούτε για τη μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού, ούτε για την εγγύηση για τους νέους. Θα τα συζητήσουμε τώρα όμως. Πρώτος, από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης του Λιθουανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Βιτάλης Ορλότ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το έτος 2013 μπορεί να χαρακτηριστεί ως σταθεροποιητική χρονιά, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι τα ε, κοινωνικά θέματα κυριαρχούν ακόμα στην Ευρώπη. Έχουμε ανεργία ε, και ε, μεγάλα προβλήματα. Το 2014 αναμένουμε μεν μια μικρή βελτίωση, αλλά η ανεργία μας ε, ανησυχεί. Ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι αποτελεσματικό εργαλείο συντονισμού των μεταρρυθμίσεων με πολυμερή εποπτεία πάρα πολύ σημαντική και παρακολούθηση. Επίσης σημαντικές είναι οι συστάσεις αναχώρα. Να είναι πιο συντονισμένες και να εφαρμόζονται. Τα αποτελέσματα και η ανάλυση αυτών θα εγγυηθούν όχι απλώς καλύτερη εποπτεία και παρακολούθηση, αλλά θα μας επιτρέπουν να διδασκόμεθα ε, μία χώρα από την άλλη. Πολύ σημαντικό είναι αυτό να έχουμε αποτελέσματα ε, για περισσότερη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων και τα κοινωνικά στοιχεία μπορούν να συμπληρώσουν τα ήδη ισχύοντα μέσα και εργαλεία που εφαρμόζουμε. Πλην όμω θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη μα ότι οι δείκτε αυτοί χωρί πρώτερη ανάλυση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω αυτόματα στοιχεία μέτρηση. Η ε, Λετωνία εξακολουθεί να αγωνίζεται ε, κατά της ε, ανεργίας, έχουμε διάφορα προβλήματα. Αυτό το καιρό καταγράφουμε την κατάσταση για να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις και να έρθουν σε αίσιο πέρας οι μεταρρυθμίσεις μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στα κοινωνικά ζητήματα και ε, στα εργασιακά. Χρειαζόμαστε βιώσιμες λύσεις, μάκρο και βράχη πρόθεσμα. Ξέρουμε ότι τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμίσεων δεν γίνονται σιτά από την αρχή. Η Λετωνία είναι μια χώρα που έχει ήδη κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως γνωρίζετε και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και να ε, υλοποιήσουμε τις συστάσεις αναχώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Από την Ιταλική Γερουσία τώρα η κυρία Μπάρμπαρα Λέτη για δύο λεπτά. Οπωσδήποτε και εμείς θα χρειαζόμασταν περισσότερη φιλοδοξία για να επιλύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας όλη την Ευρώπη. Δεν αρκεί όμως μόνο η φιλοδοξία, αλλά χρειάζεται και τόλμη. Τόλμη για να αποδεχτούμε ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές, οι πολιτικές της Τρόικας απέτυχαν. Απέτυχαν γιατί είδαμε ήδη σε όλη τη χθεσινή συζήτηση ότι δεν υπήρχαν ούτε καν θετικά αποτελέσματα στους δείκτες δείκτες που ως προς το χρέος ε, ή το έλλειμμα στο ΑΕΠ δεν έδωσαν θετικά στοιχεία. Και στην Ιταλία έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δεν υπάρχει πια περιθωριοποίησης. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε 23-24 δις άχθος των επιχειρήσεων για την κάλυψη των εργαζομένων του χρόνου προβλέπεται 34 δισεκατομμύρια αυτό το άχθος. Ε, εάν πιέζουμε διαρκώς την παραγωγική μας βάση δεν κάνουμε τίποτε. Χρειάζεται λοιπόν τόλμη και θάρρος να περιορίσουμε τη φορολογική πίεση με τρόπο αισθητό διότι ε, η νομοθεσία μας που ουσιαστικά είναι σαν προσφέρουν βοήθεια χωρίς να κάνουν κάτι μακροπρόθεσμο για το μέλλον, είναι σαν ψίχουλα στην ουσία. Ούτε στην Ιταλία λοιπόν καταφέρνουμε να προστατεύσουμε την παραγωγική μας βάση με συνθήκες εργασίας που μέχρι τώρα έδιναν σταθερότητα στην Ιταλία, διότι η Ιταλία αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα κοινωνικό ιστό, ο οποίος όμως ε, τους μεγάλους δεν τους ενδιαφέρει. Αντί να προστατεύουν και να δίνουν βοήθεια στον πολίτη, δίνουν βοήθεια στις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν προσφέρει τίποτα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η κυρία Μπάουερ από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς όλους τους ομιλητές στο βήμα. Σχετικά με τα εθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν όλες αυτές οι χώρες, δηλαδή η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Σλοβακία, εάν έχουν τέτοιο εθνικό σχέδιο και καθότι οι χώρες αυτές έχουν κάποια κοινά προβλήματα των ανθρώπων, δηλαδή χωρίς δεξιότητες και αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς, τι κάνουν για τα θέματα αυτά, διότι για παράδειγμα στη Σλοβακία η ανεργία είναι 8 φορές υψηλότερη για τους ανθρώπους ε, χωρίς ε, δεξιότητες σε σχέση με αυτούς που έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι συμβαίνει στις τρεις αυτές χώρες ε, και θα μιλήσω σλοβάκικα διότι θα ήθελα να πω κάτι στον προσκεκλημένο από τη Σλοβακία. Μιλήσατε για 70 δισεκατομμύρια την αντιμετώπιση του θέματος ε, της ανεργίας των νέων. Μάλλον κάνατε λάθος, διότι σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, 21 δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά Έτσι λοιπόν θα μπορούσατε εύκολα να λύσετε το πρόβλημα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι κάνατε λάθος ε, και όσον αφορά τις προτάσεις σας να πω ότι οι περισσότερες προτάσεις σας αποτελούν αντικείμενο ε, της αρχής της επικουρικότητας. Δεν σας εμποδίζει τίποτα να δώσετε περισσότερη να ενδυναμώσετε τις, ε, ε, τους συνεταιρισμούς και... Πρόεδρος διακόπτη την ομιλήτρια. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Τελειώσατε, τελειώσατε. Τελειώσατε. Ο Φιλίπ Κορντερή για δύο λεπτά και μετά η Βαλεντίνα Πάρης από την Ιταλική Βουλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για την εγγύηση για την νεολαία. Σας καθησυχάζω και θέλω να συγχαρώ και την Επιτροπή σας ε, που κατέστησε δυνατή αυτή την πρωτοβουλία εγγύηση για την νεολαία. Πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρώπη των πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι η γαλλική κυβέρνηση και η γαλλική εθνοσυνέλευση έχουν κινητοποιηθεί για την απασχόληση, ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων και σε επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης γιατί έχουμε εγκρίνει νόμους για το σχολείο και το πανεπιστήμιο αλλά και με ειδικά μέτρα ε, για την ε, ε, σύμβαση μεταξύ των γενεών, την θέση εργασίας για το μέλλον κτλ. Η εγγύηση για την νεολαία ισχύει από τον Οκτώβριο του 2013 στη Γαλλία. 10 είναι οι πιλωτικές περιφέρειες που δεν ταυτίζονται με τις επιλέξιμες περιφέρειες. Γι' αυτό είναι από τα προβλήματα των νομών ε, που έχουν πάνω από 25% ε, ανεργία αλλά βρίσκονται σε μη επιλέξιμες περιφέρειες. Έχουμε λοιπόν επιπλέον πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να καλυφθούν και αυτοί οι νομοί αλλά αυτό θα λειτουργήσει ως ε, ένας μαγνήτης ε, συνεργασίας του ε, κράτους, των γενικών συμβουλίων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς φορείς. Θα μπορούν λοιπόν να εντάσσονται οι νέοι στην εργασία με ε, ενεργό διαμεσολάβηση νέων και εταιριών και επιχειρήσεων. Και πάντα σε πολύ τοπικό επίπεδο γίνεται αυτή η προσπάθεια, γιατί θα πρέπει και είναι σημαντικό αυτό για μας να γίνεται όσο ε, ε, υπάρχει δυνατότητα πιο κοντά στο νέο. Είναι σημαντικό λοιπόν να ε, υπάρχει μια καθοδήγηση ευρωπαϊκή και χρηματοδότηση, αλλά η εφαρμογή να είναι ευέλικτη ε, και να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες. Ε, την Γαλλική Εθνοσυνέλευση είμαι υπεύθυνο μια έκθεση για την εργασία των νέων και με χαρά να δεχτώ τις προτάσεις των συναδέλφων που έχουν καινοτόμες ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω μέσα στο λόγο στην κυρία Βαλεντίνα Πάρης από την Ιταλική Βουλή και μετά στην Εντίτε Στρέλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και στην Ιταλία το πρόγραμμα για την εγγύηση των νέων έχει αρχίσει να εξετάζεται και έχουμε αρχίσει σε επίπεδο κοινοβουλίου τις πρώτες κινήσεις, διότι το νομοθετικό αυτό μέτρο απευθύνεται ήδη στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, διότι έχουμε το πιο νέο μέσο όρο στην ιστορία μας και τη μεγαλύτερη παρουσία γυναικών από όλη την διάρκεια ζωής της Ιταλικής Δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε συνδυασμούς και μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιο και ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουν να βρεθούν αίσθηση απασχόλησης για τους νέους και ιδίως για να καλύψουμε τις ε, διαφορές ζήτησης και προσφοράς και ζήτησης, κυρίως για τους πιο νέους. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες που προκύπτουν από τον από την, τον νόμο 92 του 2011, ιδίω για το συνταξιδοτικό μας. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να καλύψουμε αυτές, να ανατρέψουμε με αυτές που ονομάζονται στην Ιταλία εντός εισαγωγικών χρυσές συντάξεις. Λόγω αρχαιότητας και βάσει ενός νόμου ο οποίος έχει γίνει παροχημένος. Προσπαθούμε λοιπόν με το νόμο 92 να καλύψουμε τους πολίτες οι οποίοι ονομάζονται ακάλυπτοι εντός εισαγωγικών. Άνθρωποι που ξαφνικά έχασαν την ε, δουλειά τους και δεν είχαν κανένας είδος επίδομα. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής που θα αναλάβει τα ενία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα ε, ε, αναγκάσει και θα φέρει μάλλον και τον δικό μας εθνικό νομοθέτη στη θέση να καλύψει αυτό το κενό. Κενό που δεν έχει καλυφθεί λόγω του νόμου και δεν καλύπτει τις συντάξεις αυτών των ανθρώπων, πράγμα που ελπίζουμε θα γίνει στη συνέχεια. Πρόεδρος, ε, η κυρία Στρέλα τώρα για την ε, Ευρωβουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πολιτικές λιτότητας επιδεινώνουν το κοινωνικό, υποβαθμίζουν το κοινωνικό μοντέλο, καταστρέφουν τη μεσαία τάξη και αναγκάζουν τους νέους να μεταναστεύσουν. Μπορεί να έχουν πολύ ψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, αλλά παρόλα αυτά φεύγουν. Η διαρροή εγκεφάλων, λοιπόν, όπως έχει ονομαστεί, θα δυσκολεύσει την οικονομική ανάκαμψη των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, το πρόγραμμα της Τρόικας. Θα ενισχύσουν μάλιστα τις ανισότητες και τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Ο μέσος όρος νέων που δεν εργάζονται, δεν φοιτούν σε κάποιο πανεπιστήμιο, ούτε καν παρακολουθούν κάποιο κατάρτιση, είναι πάνω από 22% στις χώρες του Νότου και μόλις 11% στις χώρες του βορρά της Ευρώπης. Η εγγύηση για τους νέους είναι σημαντικότατη, αλλά δεν επιλύει όλα τα προβλήματα. Ε, Ιδίω γιατί ο προπολογισμό, τα κονδύλια που προβλέπονται από τον προπολογισμό μάλλον, είναι ανεπαρκή όπως όλοι γνωρίζουμε. Η ανεργία των νέων κοστίζει ετησίως πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Θα έφταναν μάλλον πάνω από 6 δις ευρώ, θα έφταναν 10 δις ευρώ για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια νέους από την ανεργία. Η ενεργία των νέων είναι το μείζον πρόβλημα, το μέγιστο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Είναι ακόμη σοβαρότερο από το πρόβλημα των ε, δημοσιονομικών ελλημάτων ή των κρατικών χρεών. Θα έχουμε πολύ σύντομα εκλογές το Μάιο. Ε, για Πέραν όμως της εγγύησης των νέων, τι άλλες διασφαλίσεις μπορούμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους, στη νεολαία της Ευρώπης, για να συνεχίσουν να πιστεύουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, για να κινητοποιηθούν και να ψηφίσουν στις ερχόμενες ευρωεκλογέ, για να πιστέψουν επιτέλους ότι έχουν μέλλον και στις χώρες τους και ότι δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν μετανάστες, ότι δεν χρειάζεται να φύγουν για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον εκτός της εστίας τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, ο Γκουστίν Μίζισλαβ. Πώς σας λένε, Μπασπίρτος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι εξαιρετική η προφορά σας. Έχουμε ακούσει επανειλημμένα ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στην κοινωνική πολιτική μας. Υπάρχει έλλειψη πόρων, μιλάμε για μέτρα λιτότητας και δημοσιονομική πειθαρχία. Ποια είναι η λύση όμως, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν ε, θα είναι ευχάριστο, αλλά ίσως είναι η μόνη μέθοδος. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, την απόδοση κατά την δαπάνη των πόρων μας. Υπάρχουν κάποια αποθεματικά σε κάποιους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και υπάρχει αρκετό περιθώριο ευελιξίας όσον αφορά την πιο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, ε, συμπεριλαμβανομένων των πόρων στον τομέα ε, της, ε, της κοινωνίας, των, των κοινωνικών υποθέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να έχει περισσότερο περιεχόμενο η εγγύηση που παρέχουμε με μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το σύστημα εκπαίδευσης. Η Πολωνία ακριβώς αυτό κάνει. Μεταρρυθμίζουμε το εκπαιδευτικό μας ε, σύστημα για να προσεγγίσει περισσότερο την αγορά εργασίας. Επίσης, επικεντρωνόμαστε στην διαβίου εκμάθηση και βλέπουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Φέτος, θα δούμε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις εκπαιδευτικές δαπάνες. Θα εισάγουμε τα λεγόμενα κουπόνια για ε, τις υποτροφίες για την εκπαίδευση. Οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να μετακομίσουν στα μέρη όπου υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίες. Αυτή είναι η οδός που θα ακολουθήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Λάσλο θεωρεί προτεραιότητα την βελτίωση της ελεγόμενης λευκής οικονομίας, του τομέα δηλαδή της οικονομίας που έχει να κάνει με τη φροντίδα των ελικιωμένων. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό, πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, διότι η ανεργία των νέων μπορεί να μειώνεται. Υπάρχουν προβλήματα όμως και απασχόληση σε των πιο ηλικιωμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ευχαριστώ και όλους όσοι πήραν το λόγο στη συζήτηση αυτή είτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, είτε από το Ευρωκοινοβούλιο ε, ή και τους συμμετεχόντες στο πάνελ μας. Κάπως αφαίρετα θα απαντήσω στην κυρία Μπάουερ ότι τρεις χώρες που εκπροσωπούνται στο Πρεδρείο έχουν υποβάλει τα σχέδιά τους για την υλοποίηση τη εγγύηση των νέων Απλώς, ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχουμε 160 εκατομμύρια ευρώ, 240.000 ευρώ, τα οποία μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει το ίδιο ποσό. Σε ό,τι αφορά την Ρουμανία, Πάλι έχει κατατεθεί το σχέδιο με 90 εκατομμύρια ευρώ, 99 εκατομμύρια ενώ, ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρουμανία θα πρέπει να εξαρτηθεί το ίδιο ποσό, ώστε να κινητοποιηθεί το ποσό το Ευρωπαϊκό Κονδύλι. Στη Σλοβακία το πρόγραμμα βρίσκεται υπό μελέτη, το ποσό που θα εκταμιευθεί θα είναι 67,43 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει πάλι να βρεθεί χρηματοδότηση για ένα ίδιο ποσό από τον Εθνικό Προπολογισμό. Καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά ε, περιοριστική η όλη μας προσπάθεια προκειμένου να τηρήσουμε τα όρια τα δημοσιονομικά, αλλά είμαστε όλοι στην ίδια θέση. Πρέπει να βρούμε όλοι τα μέσα μας και να σεβαστούμε τους κανόνες που θέσαμε, ιδίως για να αξιοποιήσουμε όλα αυτά που καταφέραμε με τόσο κόπο να αποσπάσουμε ως μηχανισμούς. Συγκεκριμένα τώρα για την εγγύηση των νέων. Προσπαθεί η Ευρώπη να δώσει μια απάντηση σε μια από τις μέρημνες που βρισκόνται πρώτη στις προτεραιότητες των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ να Συγχαρούμε τους ε, συμμετέχοντές μας και θα σας δώσω την ολομέλεια αμέσως. Χειροκροτήματα. Ευχαριστώ.